Spanish. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Θα, μιλήσουμε, θα μιλήσω ισπανικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλασορίζουμε ε, τους υποψηφίους για την ε, θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή να ξεκινήσω με μία σύντομη εισαγωγή. Στην αρχή αυτή τη θητεία, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου ζήτησε υποψηφιότητε για τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και καθόρισε ω ε, προθεσμία υποβολή στην 30 Σεπτεμβρίου του 2019. Στι 30 Αυγούστου του 2019 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μία ανακοίνωση για την πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητων. Δεν υπάρχει διερμηνία, τα Ιταλικά είναι στο 4. Όχι στο 7 είναι η ελληνική διερμηνία. Στις 30 Αυγούστου λοιπόν του 2019 δημοσίευθηκε στην επίσημη εφημερίδα για την ε, πρόσκληση για υποβολή υποψηφιότητων. Οι υπέβαλαν υποψηφιότητα, υποψήφοι οι οποίοι έχουν στήριξη τουλάχιστον 40 ευρωβουλευτών και είναι ε, υπήκοοι τουλάχιστον δύο κρατών μελών. Στις 23 Οκτωβρίου του 2019 ο πρόεδρος ανακοίνησε στην Ολομέλεια τις αποδεκτές υποψηφιότητες, δημοσιεύθηκε ο πλήρης κατάλογος για τους ευρωβουλευτέ οι οποίοι υποστήριξαν τους υποψηφίου. Οι υποψήφοι όλα τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για να αποδείξουν ότι πληρούν τι κατάλληλε προποθέσει. Οι υποψηφιότητε διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή μα, η οποία είναι αρμόδια για τη διοργάνωση αυτών των ακρεώσεων. Σήμερα θα ακούσουμε του υποψηφίου. Η ακρόαση είναι ανοιχτή σε όλου του ευρωβουλευτέ. Και με αλφαβητική σειρά θα ακούσουμε του εξή υποψηφίου, Ο κύριο Τζουζέπε Φορτουνάτο, η κυρία Τζούλια Λαφράνκ, ο κύριο Λίλ Σμούλσιν, η κυρία Έμιλι Οράιλι και η Σεσίλια Βίξτρομ. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάποιες πρακτικές πληροφορίες. Η ακρόαση καταρχάς ε, μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο και θα ε, μαγνητοσκοβηθούν οι παρεμβάσεις ε, των ομιλητών. Υπάρχει διερμηνία σε όλες τις επίσημες γλώσσες και θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ τους διερμηνείς, διότι σήμερα θα είναι μεγάλη μέρα. Και έχουμε αυτές τις πέντε ακροάσεις. Όπω ε, ενέκριναν οι συντονιστέ τη Επιτροπή Αναφορών, η διαδικασία θα είναι η εξή. Θα ακούσουμε του υποψηφίου με αλφαβητική σειρά. Ο καθένα θα έχει στη διάθεσή του 65 λεπτά για την ακρόαση. Κάθε υποψήφιο θα λάβει 10 λεπτά καταρχά για να παρουσιάσει την αρχική του παρέμβαση. Αυτές οι δηλώσει από εκεί και πέρα θα έχουν μια σειρά ερωταποκρίσεων. Ο πρώτο γύρο ε, θα γίνει από του συντονιστέ τη κάθε πολιτική ομάδα. και θα υπάρχει και μία απάντηση. Ένα λεπτό για την ερώτηση και τρία λεπτά για την απάντηση. Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή με το χρόνο, γιατί είναι μεγάλη μέρα, έχουμε πέντε ακροάσεις. Οι επόμενες ερωτήσεις θα είναι ένα λεπτό για την ερώτηση και ένα λεπτό για την απάντηση. Θα είναι για όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, βάσει ενός αναπλοποιημένου σύστημου, συστήματος ΔΕΟΝΤ. Το LKH2, το snd 2, ε, το Renew 1, η Πράσινη 1 η ID 1, η CR1, GUE 1 και η μία εγγεγραμμένη 1. Ε, εάν υπάρχει χρόνος θα δοθούν περαιτέρω δυνατότητες για ερωτήσεις Βέβαια της διαδικασίας Catch the Eye για 5 λεπτά. Και τέλος ο υποψήφιος θα έχει περίπου 3 λεπτά για να συνοψίσει λίγο την ε, ακρόασή του θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από όλου του ομιλητέ και για του υποψηφίου και για τα μέλη τη Επιτροπή να είμαστε λίγο πολύ τυπικοί με το χρονοδιάγραμμα. Αυτό θα κάνω εγώ σήμερα γιατί είναι μεγάλη μέρα και έχουμε πάρα πολλέ ακροάσει. Ξεκινάμε την πρώτη ακρόαση. Ο κύριο Τζουζέπε Φορτινάτο, ε, σα καλωσορίζουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ σε αυτή την ακρόαση της Επιτροπής Αναφορών, η οποία είναι ανοιχτή σε όλους τους ευρωβουλευτές για να παρουσιάσω την υποψηφιότητά μου ως ε, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Είναι η τρίτη φορά που έχω αυτή την εξαιρετική ευκαιρία σε μια ζωή στην οποία έχω επικεντρώσει ε, την επαγγελματική μου σταδιοδρομία στο προφίλ του ε, του πολίτη. Θα σας παρουσιάσω λίγο την εμπειρία μου σε τρία τμήματα. Καταρχάς, θα σας παρουσιάσω ποιος είμαι. Δεύτερον, κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και τρίτον, θα σας παρουσιάσω τις ε, γραμμές δράσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή βάσει των ε, σημαντικών δυνατοτήτων που παρέχονται, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί ελάχιστα. Είναι πολύ σημαντικό να σταθούμε στο προφίλ του συνηγόρου του πολίτη. Ο συνηγόρος του πολίτη μετατρέπει τη δυσαρέσκεια του πολίτη σε χαμόγελο. Αλλά πρέπει να μπορεί να πάει και στη ρίζα του προβλήματος. Αποφεύγοντας να υπάρχουν αντίστοιχες ε, επώδυνες καταστάσεις και δημιουργώντας και μια πιο δίκαιη δημόσια διοίκηση. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει επιτυχώς ε, τις γραφειοκρατικές αντιστάσεις, οι οποίες πολύ συχνά κρύβονται πίσω από ερμηνεία των κανόνων. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ασκήσουμε επιτυχώς τα καθήκοντα του συνηγόρου του πολίτη, πρέπει να υπάρχει μεγάλη ε, νομική δεξιότητα, κυρίως σε δημόσια ε, αξιώματα και δίνοντας κατάλληλες λύσεις. αν δεν υπάρχουν νομικέ γνώσει, ελοχεύει ο κίνδυνο όπω και στο παρελθόν να ξεκινήσουν μακρέ διαδικασίε διέρευνα χωρί να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα, δημιουργώντα ε, μια αίσθηση αδυναμία. Γι' αυτό ακριβώ και αποφάσισα να είμαι υποψήφιο για Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Δεν χρειάζεται να σα εξηγήσω γιατί θέλω να ασκήσω τα καθήκοντα του διαμεσολαβητή, δεδομένου ότι ε, αυτό κάνω και τώρα. Ήμουνα ήδη συνήγορος του πολίτη για την περιοχή της Καμπανίας από το 1999 μέχρι το 2004 και τώρα είμαι και πάλι συνήγορος του πολίτη της περιοχής της Καμπανίας από τον Ιούλιο του 2018. Ήμουνα ο πρόεδρος δύο διεθνών δικτύων ε, συνηγορών του πολίτη του Συμβουλίου του Πολίτη και του Διεθνούς Δικτύου. Από το 2015 είμαι εγγυητής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και συντονιστής του εργαστηρίου ενός ε, διεθνούς οργανισμού στον οποίο συμμετέχουν 25 εθνικές ε, αρχές ε, για προστασία των δεδομένων. Στις δραστηριότητές μου λοιπόν ήμουν επικεφαλής του νομικού και νομοθετικού γραφείου της Προεδρίας του Συμβουλίου των Υπουργών Υπήρξα διευθυντής τα ε, ε, μεταπτυχιακά προγράμματα τα οποία απευθύνονταν ε, σε επαγγελματίες και πτυχιούχους και εμβάθυνα στα βιβλία μου το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών και των εγγυήσεων για τα θέματα αυτά. έθεσα το θέμα της δημοκρατίας του πολίτη. Μια δημοκρατία στην οποία τα δικαιώματα του πολίτη εγγυώνται απόλυτα. Ο συνήγορος του πολίτη έχει το καθήκον να ε, ζητά να γίνονται σεβαστοί οι νόμοι, καταρρύπτοντας ανεπιστρεπτή την κακή διαχείριση. Να έρθω λοιπόν στα αποτελέσματά μου ως συνήγορος του πολίτη ο συνήγορος του πολίτη πρέπει να ζητά συγκεκριμένα αποτελέσματα. Όχι ένα κατάλογο των υποθέσεων και των προγραμμάτων τα οποία διαχειρίστηκε. Θα ήθελα τώρα να σας δώσω 10 παραδείγματα. Πρώτον, αμφισβήτησα τον διορισμό ατόμων που δεν κάλυπταν τις προϋποθέσεις ε, που προέβλεπαν οι ε, προκηρύξεις. Εχθές στην περιοχή της ε, Καμπανίας, ο εγγυητής για τα άτομα με αναπηρία, ο οποίος δίκαια είχε τα δικαιώματα, έλαβε τη θέση του αντικαθιστώντας κάποιον ο οποίος δεν βρισκόταν και σε αυτή τη θέση. Επίσης ζήτησαν να υπάρχουν επιτροπές εγκυώσεων για προστασία και για θέματα ισότητας των φύλων και για ε, προστασία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι Δήμοι σεβάστηκαν έτσι την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τρίτον, έκδηλες ε, παραβιάσεις της αξιοπρέπειας των γυναικών διαπιστώθηκαν σε τρεις δήμων και μέσω άμεσης παρέμβασης του συνηγόρου του πολίτη ε, υπήρξε επανόρθωση, διότι μπορούμε να έχουμε και μάχη κατά της σεξουαλικής κακοποίησης. Τέταρτο, είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για τα δάση και τις θερινές πυρκαγιές. Υποδείξαμε δημάρχους τι πρέπει να κάνουν και δώσαμε συγκεκριμένε καλές πρακτικές. Δεύτερον, κατάφερα να ε, καταρρύψω συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές ε, κατασκευές οι οποίες δημιουργούσαν φραγμούς ε, στην πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία. Επίσης, είδαμε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Εμείς θέλουμε να επιλύσουμε τις κατάλληλες ε, αντίστοιχες υποθέσεις και να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, είχαμε ως αποτέλεσμα την προληπτική ανακοίνωση ε, για τα παιδιά τα οποία ε, αποτυγχάνουν στο σχολείο πριν από τη λήξη της διαδικασίας. Ενώ ε, πριν αναλάβω συνήγορος του πολίτη είχαμε αυτοκτονίες μαθητών οι οποίοι πήραν το κακό νέο ε, ότι μένουν μεταξεταστέοι μόνο μετά την ανακοίνωση στους πίνακες στο σχολείο. Επομένω, ξεκινήσαμε μια διαδικασία υπέρ όλων. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα επίση ήταν το γεγονό ότι μειώσαμε το βάρο των βιβλίων που πρέπει να μεταφέρουν μαζί του οι μαθητέ στο σχολείο ε, μέσω μια υπόθεση ενό μαθητή και μόνον. Από τα σχολεία δίνονται έλεγχοι και σε ε, γονεί οι οποίοι είναι διαζευγμένοι, διότι στο παρελθόν δίνονταν έλεγχοι μόνο σε ζευγάρια τα οποία είναι ακόμα μαζί. Ο Στέφανο, ο νέος πατέρα, μετά από την καταγγελία που έκανε στον, Ευρωπαίο, στον ε, συνήγορο του πολίτη, επίλυσε το πρόβλημά του, αλλά και τα πρόβλημα ε, όλων των γονιών που βρίσκονται σε αντίστοιχη κατάσταση. Διαζευμένο, ο γονέας ο οποίο δεν συζεί με το παιδί του μια κοπέλα η οποία απευθύνθηκε στο συνήγορο του πολίτη για τη χρήση του κινητού τηλεφώνου για προσωπικούς λόγους στο νοσοκομείο εκτός από το γεγονός ότι τη ζήτησε συγγνώμη ε, το νοσοκομείο ε, κατάφερε να υπάρχει απαγορευτικό χρήση κινητού τηλεφώνου στα δωμάτια ε, ατόμων με σοβαρές ασθένειες που βρίσκονται στο νοσοκομείο. Επίσης, είχα και ένα πρόβλημα δραστηριότητας ως ε, ε, Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής ε, που κυρίως θέλω να εφαρμόσω κάποιες μεθόδους που έχουν ήδη εγκριθεί σε όλη τη Μεσόγειο. Να δούμε πέντε σημεία για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το άλμα ποιότητας που χρειάζεται. Καταρχάς, είναι ελάχιστες οι καταγγελίες που γίνονται στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή σχεδόν 2.200 το χρόνο, κάτι λιγότερο. Ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής λοιπόν δεν είναι γνωστός, κατά πάσα πιθανότητα διότι δεν υπάρχουν διαρθρωτικές αλλαγές ε, οι οποίες απορρέουν από τη δράση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Τα αποτελέσματα είναι η καλύτερη διαφήμιση. Δεύτερον, αυτές οι 2.200 καταγγελίες οδηγούν σε λιγότερο από 900 που είναι στην εντολή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Για τις περισσότερες καταγγελίες, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής απλώς διαβιβάζει την καταγγελία σε κάποια άλλη αρχή. Πολύ συχνά μάταια, διότι είχε ήδη αποτανθεί σε αυτές τις αρχές ε, όποιος υπέβαλε την καταγγελία πριν από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε κάθε διαδικασία και σε κάθε πράξη να δίνει και τη δυνατότητα να απευθύνεται κάποιος στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Τρίτον, δεν πρέπει να λέμε ότι τα πρότυπα της δημόσιας διοίκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλά και μόνο αυτό. Η κρίση της παρούσας Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στην ε, έκθεσή της δεν θεμολιώνεται πουθενά. Τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να ε, έχουν μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη δράση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τα ε, ευρωπαϊκέ υπηρεσίες και οργανισμούς. Πρέπει να υπάρχουν διάφορε διαδικασίε, τι οποίε πρέπει να κάνει ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πέμπτον και ολοκληρώνω, χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή με του Ευρωβουλευτέ. Δεν μπορούμε να περιοριζόμαστε μόνο σε έγγραφα και σε συναντήσει. Πρέπει να πούμε ε, με ιδιαίτερη τόλμη ότι πολύ συχνά οι ευρωβουλευτέ αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην άσκηση των καθιστών του για κάποια θέματα που διαπιστώνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία θα μπορούσε να παρέμβει συγκεκριμένα ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή πρέπει να βοηθήσει με εμπειρία, με αρμοδιότητα, με ενθουσιασμό και ανεξαρτησία για μια. Ε, ε, δημόσια διοίκηση η οποία θα βοηθά όλους να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής του. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε άλλες πτυχέ και να απαντήσω σε ερωτήσεις γενικότερα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φορτουνάτο, κύριε υποψήφιε. Θα ξεκινήσουμε με τους συντονιστέ. Και πρώτα απ' όλα δίνω τον λόγο στον κύριο Πίτερ Γιάρ, ένα λεπτό συντονιστή του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Φορτουνάτο για την ε, παρουσίαση σας. Έχω μια σύντομη ερώτηση. Πώς βλέπετε τη συνεργασία μεταξύ περιφερειακών ε, ε, συνηγόρων του πολίτη με τον Ευρωπαίο συνήγορο και πώς ορίζετε τα όρια της αρμοδιότητάς σας, του έργου σας ως Ευρωπαίου δημοσιολόγητη; Πώς θα διακρίνετε δηλαδή που τελειώνει η δική σας δικαιοδοσία. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Και ευχαριστώ που έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε πέντε υποψηφίους, ε, κάτι που προσδίδει περισσότερη αγωνία σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Φορτουνάτο, παρακαλώ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Πρόκειται για κεντρικό ζήτημα, αυτό δηλαδή της ε, συνεργασίας, έτσι ώστε ο ένας να μάθει και από τον άλλον. Είναι ε, πολλοί ε, οι διαμεσολαβητές, ε, με όποιο όνομα και αν έχουν, συνήγοροι του πολίτη, ε, τα κτλ, ε, που εν τέλει είναι οι φίλοι του πολίτη. Και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει η ενιαία θηρίδα των συνηγόρων του πολίτη και μετά το International Ombudsman που αφορά τους διαμεσολαβητές σε όλο τον κόσμο. Το πρόβλημα των διαμεσολαβητών είναι ακριβώς αυτό το θέμα της αντίθεσης προς ε, την δημόσια διοίκηση και της αλλαγής ε, των κανόνων του παιχνιδιού. Αυτή είναι ε, η συζήτηση. Αυτό είναι ο διάλογος που πρέπει να έχουμε έτσι ώστε να μάθουμε ο ένας από τον άλλον. Και νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε αφήγημα ε, ε, σύμφωνα με το οποίο δηλαδή ε, ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής θα πρέπει να αποτελέσει μοντέλο, πρότυπο που θα ακολουθούν και οι άλλοι. Και εμείς μπορούμε να μάθουμε από τους άλλους έτσι ώστε να μπορέσουμε να ακούμε προσεκτικά και να δίνουμε λύσεις και ικανοποίηση τελική εις τον πολίτη. Θα πρέπει πάντοτε βέβαια να εγγυόμαστε ε, την ανεξαρτησία μας και την ικανότητα να λύνουμε ε, δίκαια τα προβλήματα. Γιατί διαφορετικά ε, εάν δημιουργήσουμε αυτήν την εικόνα ενός διαμεσολαβητή στον οποίον προσφεύγει κανείς και ο οποίος δεν καταφέρνει να λύσει τα προβλήματα τότε θα δημιουργηθεί το αίσθημα της αδυναμίας του διαμεσολαβητή. Αυτό ήθελα να πω εγώ. Και κυρίως το ότι ο ένας πρέπει να μάθει από τον άλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κριστίνα Μαέστρε από τους Σοσιαλιστές. Ε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Φορτουνάτο ε, για την παρουσία σας εδώ στην Ακρόαση και ευχαριστούμε για τις ε, θέσεις σας. σας άκουσα ε, με προσοχή, διάβασα την εμπειρία σας, διάβασα το βιογραφικό σας, ε, τις διάφορες θέσεις ευθύνης που είχατε ε, όχι μονάχα σαν συνήγορος του πολίτη στην καμπανία αλλά και άλλες θέσεις που είχατε. Αναφερθήκατε στην εσωτερική διαβούλευση, στην ενίσχυση του διαμεσολαβητή και της εικόνας του διαμεσολαβητή. Ε, αναφερθήκατε επίσης ε, στον μικρό αριθμό των καταγγελιών που φτάνουν περίπου στις 2.000 ε, και είπατε ότι πρέπει οπωσδήποτε να εργαστούμε έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει των πολιτών. Συμφωνούμε με εσά ότι θα πρέπει να προσεγγίσουν τα ευρωπαϊκά όργανα εις τους, τους πολίτες. Ποια είναι τα σχέδιά σας, το πρόγραμμά σας έτσι ώστε να μην ε, ζούμε πραγματικά σε ένα είδος ε, ε, φούσκας ας πούμε αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. Πώς θα προσεγγίσουν όντως τα όργανα τους πολίτες. Δεν, ξέρω εάν μπορείτε να αντιλήσετε εμπειρίες από τις προηγούμενες θέσεις σας, αλλά με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό και πώς θα κινηθείτε έτσι ώστε να ενισχύσετε την εικόνα του διαμεσολαβητή. Κύριε Φορτουνάτο. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Μικρόφωνο. Κοιτάξτε, ο συνήγορο του πολίτη, ο διαμεσολαβητή δηλαδή, είναι ο φίλο του πολίτη. Ο φίλο ο οποίο θα σταθεί στο πλάι του και θα λύσει τη δυσκολία. Ε, εμείς ε, θέλουμε να πηγαίνει κανεί στον συνήγορο του πολίτη όπως θα πήγαινε ε, σε ένα νοσοκομείο εάν έχει πρόβλημα. Ε, και η λειτουργία του συνηγόρου του πολίτη είναι ακριβώς το συγκεκριμένο αποτέλεσμα να μπορέσει να πει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση λύθηκε το πρόβλημα. Κυρίως, κυρίως όμως ε, όχι απλώς να πει ότι λύθηκε το θέμα, αλλά ότι βάσει του συγκεκριμένου ζητήματος που λύθηκε θα δημιουργηθούν, θα θεσπιστούν νέοι κανόνες. Εμείς ε, ικανοποιούμε τον καταγγέλλοντα, αλλά φτάνουμε και στη ρίζα του προβλήματος έτσι ώστε τέτοιου είδους προβλήματα να μην ξαναπαρουσιαστούν. Μόνο με τον τρόπο αυτό ε, καταπολεμάμε την κακή διοίκηση. Εδώ ε, βεβαίως πρέπει να είναι σαφές ε, ότι θα πρέπει να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα, θα πρέπει να γίνουν παρουσίες ε, στο διαδίκτυο, να γίνουν διασκέψεις, να γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως πρέπει πρώτα να υπάρχουν αποτελέσματα. Η παρουσία του συνηγόρου του πολίτη θα πρέπει να σηματοδοτεί μια διαφορετική σχέση του πολίτη με το κράτος, με τη διοίκηση και γι' αυτό πιστεύω ότι ο διαμεσολαβητής για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερα και προηγουμένως, γιατί υπάρχουν και κοινοβουλευτικά ερωτήματα τα οποία αφορούν πολύ σοβαρά προβλήματα, ε, τα οποία όμως δεν καταφέρνουμε να, να λύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ομάδα Renew, η κυρία Τόμ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα και για τις απαντήσεις που δώσατε. Πριν τη συνεδρίαση αυτή είχαμε συνεδρίαση συντονιστών και για άλλη μια φορά συζητήσαμε τις ε, γεωγραφικές ανισορροπίες, τις ε, διαμαρτυρίες. Αν δούμε μια μελέτη του Ευρωβαρόμετρου που έγινε τον Μάιο του 2019, το πώς κατανοούν οι πολίτες ε, διαφόρων κρατών τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ, διαφέρει πολύ Στι ερωτήσει, όπω αν υπάρχουν ε, εθνοτικέ διακρίσει στη χώρα σα, το 76% των πολιτών στην Ολλανδία θεωρούσαν ότι υπήρξε μεγάλο πρόβλημα, αλλά στην Λετωνία που πραγματικά υπάρχουν προβλήματα σε εθνοτικέ διακρίσει, μόνο το 25% των πολιτών ε, το πίστευε αυτό. Άρα το ερώτημά μου είναι αν βλέπετε κάποια λύση. Για να πλησιάσετε τον κόσμο, να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο πώς μπορούν να υποστηρίξουν τον εαυτό τους, να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Και επίση αν μπορείτε να εξασφαλίσετε κάποια ισορροπία γιατί υπάρχουν ε, κράτη-μέλη που υπάρχουν πολύ δραστήριοι πολίτες και μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά σε άλλες δεν υπάρχει κάτι ανάλογο. Δεν θα τις ε, κατονομάσω τις χώρες αυτές, αλλά πείτε μου ποια είναι η άποψη σας επί αυτού. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να καταπολεμηθούν ε, οι διακρίσεις. Θα πρέπει να δοθεί σε καθέναν την δυνατότητα ε, να εκφράζεται ελεύθερα και να προασπίζεται την κεραιότητα ε, των ατόμων και την αξιοπρέπεια των ατόμων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σε σχέση με τα δικαιώματα. Ο διαμεσολαβητής είναι ο δεύτερος συνήγορος του πολίτη. Ο πρώτος συνήγορος του πολίτη πρέπει να είναι ο ίδιος ο πολίτης που δεν πρέπει να ε, δέχεται ούτε ο ίδιος να υφίσταται διακριτική μεταχείριση, ούτε ε, να μεταχειρίζεται με διακριτικό τρόπο, διαφορετικό τρόπο τους άλλους και ε, νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο ε, και ο διαμεσολαβητής ε, θα μπορέσει να παίξει τον κυρίαρχο ρόλο του που είναι αυτό της προώθησης της δικαιοσύνης. Γιατί ο διαμεσολαβητής αυτό κάνει, προωθεί τη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Όουκεν από τους Πράσινους παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Είμαι λίγο έκπληκτη που κατηγορείται την ε, τρέχουσα διαμεσολαβήτρια ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της, γιατί είναι θέμα νομοθεσίας. Δεν μπορεί να διαχειριστεί καταστάσεις οι οποίες αφορούν τους εθνικούς διαμεσολαβητές. Είναι δικό τους θέμα. Με εκπλήσει λοιπόν αυτό αλλά φαίνεται ότι είστε πολύ επικριτικός για το πώς έχουν διαχειριστεί καταστάσεις προηγούμενοι διαμεσολαβητές. Το προνόμιο που έχουν για τις ε, εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Αυτό συμπεριλαμβάνεται στην θήκη του 2008. Πώς το βλέπετε εσείς το θέμα αυτό για τις ε, εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτό το προνόμιό σας. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί πρόκειται για πολύ ουσιώδες θέμα. Εγώ σέβομαι ε, την δράση της Έμιλι ε, Ρέιλι, η οποία έδωσε πολύ από τον εαυτό της σε όλες τις ε, ε, συζητήσεις. Αλλά ε, έχουμε και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχουμε τρεις εκστρατείες, οι οποίες όμως στην ουσία δεν έδωσαν κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα και ακριβώς δημιουργήθηκε μία έννοια αδυναμίας. Η διαμεσολαβητής Ορέλη αναφέρθηκε στον Μπαρόσο, δεν άλλαξε όμως τίποτα. Επίσης, ε, η Ευρωπαία Διαμεσολαβητής αναφερθήκε στον ε, Σέλμαρ ε, σχετικά με τα θέματα αυτά τα οποία ανέμειξαν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τίποτα δεν έγινε. Επίσης, ε, η Μεσολαβητής μίλησε για τον ε, πρόεδρο Ντράγκη, πρόεδρο της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και μέλος της ομάδας των 30. Δεν έγινε όμως κάτι και γι' αυτό. Γνωρίζω ότι και στα θέματα αυτά υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει και μπορεί να ε, ε, λύσει ή να αναλάβει ο διαμεσολαβητής. Εν πάση περιπτώσει όμως, ο προπονητής κρίνεται από τα αποτελέσματα της ομάδας του. Ε, γι' αυτό ακριβώς εγώ σας είπα ότι... έχω πετύχει συγκεκριμένα πράγματα στην δικιά μου περιφέρεια και ας πούμε χθες ακόμα ε, εγώ κίνησα το θέμα του εγγυητή των ανθρώπων με αναπηρία και άλλαξα τον άνθρωπο ο οποίος θα έπαιρνε την θέση αυτή. Η κυρία Ορέλη είναι δημοσιογράφος, ε, ε, είναι πολύ καλή δημοσιογράφος, κάνει ερευνητική δημοσιογραφία με, μεγάλη, έτσι, με μεγάλο αποτέλεσμα όσον αφορά τη δημοσιότητα. Αναφέρθηκα λοιπόν σε αυτές τις τρεις εκστρατείες που πήραν μεγάλη μεγάλη δημοσιότητα, αλλά καμία από αυτέ ε, δεν οδήγησε σε κάποιο συγκεκριμένο πράγμα. Αποτέλεσμα, ε, ο πολίτη όμω ε, λέει έρχομαι σε σένα γιατί δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι υπάρχει, υπάρχουν εξουσίε και προνόμια του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή αυτές τις εξουσίες και αυτά τα προνόμια θα πρέπει να τα υλοποιήσουμε σε βάθος, να δούμε πού υπάρχουν παραβιάσεις και να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλες τις εξουσίες, τα προνόμια, τα δικαιώματα που έχουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε αποτελέσματα. Εμείς δεν χρειαζόμαστε μονάχα κάποιον ο οποίος θα λέει αυτά δεν λειτουργούν καλά ή τα άλλα δεν λειτουργούν καλά. Στην Ευρώπη χρειαζόμαστε έναν Ευρωπαίο διαμεσολαβητή που να λύνει τα προβλήματα του πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λοτόφσκι παρακαλώ. E, Καλημέρα σας. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου και έχω τρεις ερωτήσεις. Σε ποιους τομείς υπάρχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων ε, στους, στα θεσμικά όργανα. Δεύτερον, θα θέλατε να φέρετε πιο κοντά στους πολίτες τη διαδικασία ε, διαπραγμάτευσης ε, νομοθετικών πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίση ε, η διαδικασία των τριμερών διαλόγων θεωρείται ότι είναι αρκετά διαφανή για του Ευρωπαίου πολίτε και αν όχι, πώ θα θέλετε να το αλλάξετε αυτό. Σα ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ο γητής της διαφάνειας με εξαίρεση κάποιες συγκεκριμένες ε, υποθέσεις ε, προστασίας ε, αξιών και προστασίας δεδομένων. Η βασική αρχή όμως η οποία θα πρέπει να διέπει όλη την δημόσια διοίκηση της Ευρώπης είναι η αρχή της διαφάνειας. Και ο εγώ συνήγορο του πολίτη πολύ συχνά ασχολούμαι με την πρόσβαση στι νομικές πράξει. Ε, πολλέ φορέ ε, οι δημόσιες διοικήσεις δεν δίνουν τις διάφορες πράξεις ε, βρίσκοντας διάφορες δικαιολογίε. Από την έκθεσή μου σε πολλέ περιπτώσεις έχω καταφέρει να δοθούν οι διάφορες πράξεις στου πολίτε. και αυτό πολύ συχνά ε, δεν βρίσκονται στο σκοτάδι μόνο οι Ευρωπαίοι πολίτε, αλλά ακόμα και οι Ευρωπαίοι βουλευτές. Δηλαδή, εμεί σα ψηφίζουμε, είστε οι αιρετοί του λαού, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα τη ευρωπαϊκή διοίκηση, το οποίο είναι εκτό οποιασδήποτε πραγματικής απέτηση διαφάνεια. Όπω για παράδειγμα οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί και υπηρεσίε, στου οποίου γνωρίζουμε ελάχιστα για το τι γίνονται και η διαφάνεια δεν είναι και ίδιον αυτών των οργανισμών και των υπηρεσιών. Εσεί, λοιπόν ως ευρωβουλευτές θα πρέπει ε, να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τέτοιο εργαλείο. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε και θέματα που αφορούν την πρόσβαση όχι μόνο στις ε, τελικές ε, διατάξεις, αλλά και τη δυνατότητα της συμμετοχής των πολιτών στην όλη διαδικασία. Τη δυνατότητα δηλαδή να μπορεί ο καθένας να ε, γνωρίζει πώς συμμετείχε ο κάθε ενδιαφερόμενος. Και εδώ έρχομαι και στο τελευταίο σκέλος της ερώτησης που μου θέσατε. Ευχαριστώ πολύ. Από την ΚΟΕ δεν βλέπω εδώ τον κύριο Γεωργούλη και δεν βλέπω και κάποιον άλλον από την ΚΟΕ. Να περάσουμε λοιπόν στον κύριο Βίντσε από το ΕΛΚ. Βίντς. Ευχαριστώ. Αγαπητέ υποψήφοι, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ τεχνική, κατά την άποψή μου. Ας προσπαθήσουμε να μιλήσουμε τώρα για έναν τομέα που είναι πολύ σημαντικός για αυτή την Επιτροπή, γιατί υποστηρίζουμε όχι μόνο τους αναφέροντες, αλλά προσπαθούμε να υποστηρίξουμε όσο περισσότερα γίνεται και την καλύτερη συμμετοχική δημοκρατία συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλειών των πολιτών. Υπάρχει ένας νέος ε, κανονισμός που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Το γραφείο του διαμεσολαβητή έχει πολύ σημαντικό ρόλο και μια επιτροπή πολιτών συνάντησε διοικητικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς βλέπετε το ρόλο του διαμεσολαβητή στην στήριξη των πρωτοβουλειών των πολιτών και πώς μπορείτε να συνεισφέρετε περισσότερο ε, σε αυτό το θέμα υπέρ των πολιτών. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι συμβάλλω συνεχώς στη δραστηριότητά μου στο θέμα της συμμετοχής. Για παράδειγμα, στην Ιταλία στα πάρκα πρέπει να υπάρχει κανονισμός για τη συμμετοχή, ώστε να μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν σε όλα όσα αφορούν ε, τα το περιβάλλον. Τα πάρκα δεν είχαν τέτοιο κανονισμό και εγώ απευθύνθηκα στους προέδρους ε, των ε, πάρκων και ζήτησα και από τους υπουργούς ε, να διαλύσει το Διοικητικό Συμβούλιο, διότι το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ε, δεν τηρούσε τους κανόνες, δεν μπορούσε να παραμείνει. Και ενώπιον αυτής της απειλής ε, ε, κατέθεσαν και διαδικασίες για συμμετοχή των πολιτών. Το ίδιο έκανε και για τους Δήμους. Στους Δήμους δεν υπήρχε κανονισμός για τη συμμετοχή, επομένως δεν υπήρχε εγγύηση της αρχής της κυριαρχίας του λαού και της συμμετοχής του πολίτη. Και ε, εγώ τους αμφισβήτησα και ενέκριναν κανονισμό μόνο μετά από από την αμφισβήτηση του συνηγόρου του πολίτη. Δηλαδή, πολλές φορές υπάρχουν αντιστάσεις από κάποιους ε, γραφειοκράτες ε, και από κάποιους ε, διοικητικούς υπαλλήλου, οι οποίοι δεν θέλουν να συμμετέχει ο πολίτης στο δημόσιο βίο. Και αυτό που λέω συχνά είναι ανοίξτε τις πόρτες στους πολίτες. Ο κανονισμός ο οποίος εγκρίθηκε μετά από πρωτοβουλία του συνηγόρου του πολίτη σε ένα δήμο στο Τσασάνο είναι κανονισμός για την συμμετοχή, την ιδιαίτερα προηγμένη συμμετοχή άλλωστε. Διότι προβλέπει καταρχάς ένα κώδικα διοντολογίας για τους δημοσιογράφους δημόσιους λειτουργούς ε, και επομένως ε, υπόκεινται και σε ε, ε, διοικητική εξέταση και μπορεί ο πολίτης να ζητήσει πραγματικά να τηρηθεί ο κανονισμός. Ο διαμεσολαβητής λοιπόν πρέπει να είναι ο εγγυητής, ο προστάτης του πολίτη και να μπορεί να προσφύγει για τα δικαιώματά του. Αυτά λοιπόν εγκρίθηκαν από το συνόργο του πολίτη γιατί ο Δήμος δεν φρόντιζε να προβλέψει καταλήλως χρησιμοποιώντας ε, την Ιταλική νομοθεσία η οποία ούτως ή άλλως ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο προέλευε και ε, συμμετοχή ε, και κοινωνική συμμετοχή. Προβλέπεται λοιπόν συμμετοχή στον προπολογισμό και σε κοινωνικά ζητήματα και ε, κάποια άλλους, άλλες δυνατότητες, για παράδειγμα ένα ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο, ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο να συμμετέχουν και οι υπεύθυνοι της κοινωνίας των πολιτών, όχι μόνο οι αιρετοί. Αυτό δεν είναι μόνο απλώς μία επιβεβαίωση μιας αρχής, είναι ένας κανονισμός ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί και ο οποίος φυσικά θα μπορούσε να αποτελέσει και ε, οδηγό για να συνεχίσουμε να ανοίγουμε τις πόρτες στους πολίτες. Και τώρα ε, κανονικά ε, ήταν η σειρά των σοσιαλιστών. Δεν συμμετέχει, ο, δεν είναι εδώ ο κύριος Άλεξ, ο κύριος Άμενιξ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Υπάρχουν ησυχίες στο δημόσιο τομέα. Ο ρόλος σας ως διαμεσολαβητή είναι να διερευνήσετε την κακοδιοίκηση σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς με την έλλειψη εμπιστοσύνης που αισθάνονται οι πολίτε έναντι των θεσμών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Πώς ε, προτίθεστε να μειώσετε το κενό μεταξύ πολιτών, το χάσμα μεταξύ πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκεκριμένα. Ε, Κοιτάξτε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πραγματικά ένα εργαλείο ε, έτσι ώστε ο να μπορούν να συζητούν ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτες και ο ε, διαμεσολαβητής ε, πραγματικά είναι μια τέτοια εικόνα που δημιουργήθηκε πριν από δύο αιώνες στην Σουηδία. Ένας πραγματικός αρμόδιος διοικητικός διαμεσολαβητής για να δώσει και φωνή στον πολίτη που συχνά δεν έχει φωνή. Πολύ συχνά ο πολίτης λέει πράγματα σωστά αλλά δεν μπορεί να ακουστεί η φωνή του. Ε, και ο διαμεσολαβητής είναι το μεγάφωνο μέσω του οποίου θα ακουστεί η φωνή του πολίτη. Ε, και με τον τρόπο αυτό οικοδομείται εμπιστοσύνη. Γιατί στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, το βασικό θέμα είναι ακριβώς αυτό της σχέσεις ανάμεσα στον πολίτη εκλογέα ε, και το, τους πολιτικούς. Δηλαδή ε, οι πολίτες έχουν συχνά την εντύπωση ότι οι πολιτικοί έρχονται, ε, ζητούν την ψήφο και μετά ξανάρχονται, γίνονται οι εκλογές, ξανάρχονται μετά από τέσσερα χρόνια. Ενώ ο διαμεσολαβητής ε, είναι παρόν διαρκώς. Η κυρία Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής ασκεί τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο, αλλά έχει στενή σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το είπατε σε προηγούμενη απάντηση, η Ευρωπαϊκή Διοίκηση ε, θα πρέπει να ε, ανταποκρίνεται ε, στις ε, απαιτήσεις διαφάνειας. Έχουν γίνει κάποιες προτάσεις, αλλά βεβαίως πρέπει να πω ότι υπάρχουν καταγγελίες και προσφυγές και για το Κοινοβούλιο. Κατά την άποψή σας, ποια είναι τα προβλήματα, τα διοικητικά τα οποία συνδέονται με το Κοινοβούλιο και πώς μπορούν να αρθούν αυτά τα προβλήματα. Κοιτάξτε, εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες ψηφίζουμε ε, τους Ευρωπαίους πολιτικούς ε, και ε, ε, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο οίκημα το οποίο σας ε, βοηθάει έτσι ώστε να ασκήσετε το καθήκον σας αυτό της εκπροσώπησης των Ευρωπαίων πολιτών. Οποιαδήποτε λοιπόν λειτουργία έτσι πρέπει από αυτή την οπτική γωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζετε εσείς ως ε, εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών θα πρέπει ε, να κινηθείτε έτσι ώστε όλη η νομοθεσία και όλοι οι διοικητικοί κανόνες να έχουν σαν γνώμονα την προστασία του πολίτη. Τότε θα έχουμε πετύχει. Εάν όμως εσείς ε, ως πολίτες, ως Ευρωπαίοι βουλευτές ε, δεν μπορείτε να κάνετε κάτι ε, και κατά κάποιο τρόπο αισθάνεστε εφημωμένοι ε, τότε και ο πολίτης πραγματικά δεν θα μπορεί να αισθανθεί ότι μπορεί να βρει το δίκιο του. γι' αυτό λέω ότι κάθε καταγγελία θα πρέπει να ελέγχεται σε βάθος. Ευχαριστώ κύριε Σκόζα. Köszönöm Είμαι πολύ χαρούμενος που στη σημερινή ακρόαση και βλέποντας το βιογραφικό σας παρατηρώ ότι έχετε κάνει πολλές προτάσεις στο παρελθόν και γι' αυτό ε, έχω την εξή σε σχέση με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς θα εφαρμόσετε τους κανόνες που τα αφορούν θα επεκτείνετε το πλαίσιο ή θα ακολουθήσετε κατά γράμμα τους κανόνες. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα άτομα με αναπηρία. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία, οπότε είναι πολύ κατάλληλη η στιγμή να θέσω αυτό το ερώτημα. Δυστυχώς εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν γίνει πολύ λίγα αιτήματα στο διαμεσολαβητή από άτομα με αναπηρία και πιστεύω ότι ο ένας λόγος γι' αυτό είναι ότι δύσκολο για τα άτομα αυτά να έχουν πρόσβαση Άρα σας ρωτάω πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό στο μέλλον. Ευχαριστώ. Το πρώτο ερώτημα αφορά τις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Εγώ πιστεύω ότι και επί τη βάση του υφιστάμενου κανονικού, κανονισμού ε, προβλέπονται ε, ε, δικαιώματα και προνόμια τα οποία μπορούν να επιτρέψουν στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή να μελετήσει το θέμα επί της βάσεως της δυνατότητας συγκεκριμένου αποτελέσματος. Μπορούν να εξεταστούν και άλλες δυνατότητες, δηλαδή να δοθεί στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή μια δυνατότητα ε, βάσει της οποίας εάν ε, κάποια γραφειοκρατική αρχή ε, δεν συμμορφώνεται να έχει τη δυνατότητα το διαμεσολαβητής να λύσει το πρόβλημα χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσουν δικαστικές διαδικασίες. Αυτό είναι πολύ καλό και για τους πολίτες που δεν έχουν και τόσα χρήματα έτσι ώστε να λύσουν ε, νομικά το θέμα. Και ε, υπάρχει βέβαια το άλλο ζήτημα, το ζήτημα ε, των ανθρώπων με αναπηρία. Εκεί πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόζονται όλες, όλα τα νομοθετικά κείμενα ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αρθούν ε, πολλοί αρχιτεκτονικοί φραγμοί σε ε, πολλές κοινότητες. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται πάντα ο νόμος και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής οπωσδήποτε θα είναι πάντα στο πλευρό όλων των Ευρωπαίων πολιτών που χρειάζονται προστασία. Να σας υπενθυμίσω ότι τώρα πια έχουμε περάσει ε, στις ερωτήσεις και απαντήσεις ενός λεπτού. S&D Άμεριξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Δεύτερο ερώτημα. Για να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση των απόψεών σας, θα ήθελα να σας ρωτήσω μια μικρή αλλά πολύ σημαντική για όλους μας ερώτηση. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι μεγαλύτερος από το να είναι νομικός διαμεσολαβητής. Ποιοι θέλετε είναι συγκεκριμένοι στόχοι που θα θέλετε να πετύχετε κατά τη διάρκεια της θητής σας και ποιοι θα είναι οι τρεις τομείς εργασίας στους οποίους θα ε, θέλετε να ε, αποδώσετε. Sono η στόχοι του συνηγόρου του πολίτη είναι η δημόσια διοίκηση να γίνει πιο ευγενική, πιο αποτελεσματική, πιο ανθρώπινη, πιο αποδοτική και πιο δίκαιη. Ο συνήγορος του πολίτη πρέπει να απαντά σε ένα απλό ερώτημα. Έχω κάνει τη, δική, τη δημόσια δίκη πιο δίκαιη, πιο αποτελεσματική, πιο υγιή. Και εδώ υπάρχει ένα πρόγραμμα πρέπει οποιοδήποτε ερώτημα να το απαντούμε αναρωτιόμενοι πώς μπορούμε να φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί. Το θέμα λοιπόν είναι ο πολίτης να είναι σε θέση να νιώσει ότι η δημόσια διοίκηση είναι στην υπηρεσία του. Γιατί συμβαίνει σε εμά του ανθρώπου κάτι πάρα πολύ περίεργο. Υπό την έννοια ότι δημιουργούμε τις δημόσιες αρχές, τους δήμους, τις επαρχίες και τις περιφέρειες και τελικά φαίνεται να είναι όλα μηχανισμοί που είναι εκτός από τον πολίτη. Ενώ ο διαμεσολαβητής είναι αυτός ο οποίος βοηθά τον πολίτη και παρεμβαίνει ανταυτού. Υπενθυμίζει πάντα σε κάθε δημόσια εξισία ότι είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Η πιο συγκεκριμένη μέθοδος που γίνεται σε κάποια ε, περίπτωση είναι αυτή η οποία θα πρέπει να μετατρέψουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι το άλμα ποιότητας που πρέπει να έχει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Η κυρία Στάνοκα. Ευχαριστώ κύριε Φορτουνάτο. Για την παρουσία σας δύο ερωτήσεις. Πρώτον, κατηγορήστε την κυρία Μιλή Ρέιλι ότι δεν ήταν πολύ δραστήρια στην θέση της και γι' αυτό υπήρξαν πολύ λίγα αιτήματα στο διαμεσολαβητή. Πόσα αιτήματα είχατε εσείς ως ε, περιφερειακός διαμεσολαβητής και ποιος ήταν ε, ο δικός σας ρόλος. Είχατε περισσότερα αιτήματα αναλογικά με αυτά που είχε η Ευρωπαϊκή Διαμεσολαβητής και δεύτερον. Όσον αφορά τη διαφάνεια, είπατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει επιρροή στους στα θεσμικά όργανα για να υπάρχει διαφάνεια. Αν όμως το Συμβούλιο απορρίψει αυτή την πρόταση, πώς θα ληφθεί η απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι δύσκολο να επηρεάσουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Ναι, οι ερωτήσει είναι δύο. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, εγώ ασχολούμαι με χιλιάδες προσφυγές, ε, υποδείξεις, και μόνο βρισκόμενο σε μια μικρή περιφέρεια, διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τόσες πολλές χώρες ο αριθμός των 2.200 καταγγελιών είναι πάρα πολύ χαμηλός, διότι Μόνο στην καμπάνια εγώ έχω 4.000 με 5.000 καταγγελίες από πολίτες που έχουν διάφορα προβλήματα ε, διαφορετικής φύση ο καθένα. Όσον αφορά του ευρωβουλευτέ, είπα ότι ο, ο συνήγορος του πολίτη και σε αυτή τη φάση στο οικοδόμημα τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο συνήγορο του πολίτη του ευρωβουλευτή. Διότι υπάρχει ένα 90% της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο διαφεύγει από τους ερετούς εκπροσώπους του πολίτη. Ο πολίτης καλείται να αποκαλεί εσάς εκπροσώπους του πολίτη και δεν είναι δυνατόν εσείς να μην έχετε δυνατότητα παρέμβαση. Εγώ βλέπω μια αλλαγή εδώ. Θεωρώ ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα πρέπει να σας βοηθά και το βλέπω αυτό ξεκινώντας από τα ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών που διάβασα που διαπιστώνουν πολλές περιπτώσεις κακοδιαχείρισης δημόσιας διοίκησης οι οποίες δυστυχώς συνδέονται και αυτές με ένα γραφειοκρατικό παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχει μια ερώτηση, μια απάντηση και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Αν μπορέσουμε όμως να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταγγελίες και θέσουμε προληπτικά το θέμα της απάντησης, μπορούμε να δούμε αν έχουμε τις εξουσίες για να επιλύσουμε το ζήτημα. Αλλιώς είναι κάτι αρνητικό. Δημιουργείται μια απογοήτευση. Αν ξεκινήσει μια διαδικασία η οποία τελικά έχει αρνητικό αποτέλεσμα, είναι κακή διαφήμιση για τα θεσμικά όργανα και αυτό φυσικά δεν είναι καλό και για κανέναν. Ευχαριστώ. Ο κύριο Στρακανέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χωρί μικρόφωνο και ο κύριο Στρακανέλη. Micro, micro. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τη σκέψη σας και διάβασα και το βιογραφικό σας όπως έκανα και με του υπόλοιπου υποψηφίου. Το καθήκον του Ευρωπαίου ε, βουλευτή είναι να επιλέξει τον υποψήφιο ο οποίος θα μπορέσει να εγγύθει την αρμοδιότητα και την ανεξαρτησία στην άσκηση των καθηκόντων του ως Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Δηλαδή όταν θα ψηφίσουμε εμεί στο Στρασβούργο δεν θα διαλέξουμε εάν ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή μπορεί να εκπροσωπήσει το τάδε το δίνα συμφέρον, αλλά αν μπορεί να ε, απαντήσει στι απαιτήσει των πολιτών. Για να απαντήσω λοιπόν ε, σε αυτό που μόλις είπατε, θεωρείτε εσείς ότι έχετε τις αρμοδιότητες. Θέλετε να μας εξηγήσετε και γιατί θεωρείτε ότι είναι δική σας αρμοδιότητα στο βιογραφικό σας, οι δραστηριότητε σας και το πρόγραμμά σας, όπως μας παρουσιάσατε εδώ, απαντώντας τις ερωτήσεις των συναδέλφων, είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει να προτιμήσουμε εμείς σε σχέση με τους άλλους υποψηφίους. Τι είναι αυτό που σας διακρίνει λοιπόν με βάση τα όσα κάνατε και τα όσα είπατε σε σχέση με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο και πάλι. Έχω άρτια νομική κατάρτιση όσον αφορά την νομοθεσία διότι πρέπει να δίνουμε απαντήσεις ε, σεβόμενοι και τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα διεύρυνα και τι γνώσει μου όσον αφορά τη συγκεκριμένη αλλαγή εντό των διαδικασιών. Για παράδειγμα, κάποιο, ο οποίο μπορεί να έχει νομική κατάρτιση, ε, αλλά είναι δικαστή. είναι σε θέση να εκδώσει μια απόφαση, να επιβεβαιώσει καν κάποιο έχει δίκιο ή άδικο, αλλά είναι τελείω διαφορετικό το να είναι κάποιο διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητή πρέπει να προσεγγίζει το πολίτη για την επίλυση του προβλήματός τους. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι εύκολη δουλειά, να ε, μετατρέψουμε τη δυστυχία σε χαμόγελο. Μπορείτε εσείς να κάνετε το γιατρό, όταν, θα βάζετε κάποιον να κάνει το γιατρό όταν δεν έχει τις δεξιότητες, θα βάζετε κάποιον ε, να κάνει κάποια δουλειά που δεν έχει τις συγκεκριμένες δεξιότητες. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με καλή βούληση, αλλά ποτέ δεν μπορεί να δώσουν αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που μπορεί να δώσει ο διαμεσολαβητής, εφαρμόζοντας πλήρως την νομοθεσία και δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε διαδικασία να επιληθεί το πρόβλημα, να υπάρχει η τεχνική, η μέθοδος και η δυνατότητα να επιλύσει κάποιος θετικά ε, μια υπόθεση. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, κανονικά είναι η σειρά του κυρίου Μακάρθη από την ΚΟΕ, ούτε και τον κύριο Μάριο Φουρόρα όμως βλέπω. Επομένως εδώ ολοκληρώνεται αυτή η ακρόαση. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος το λόγο στο Catch ή μπορεί να το κάνει κάλλιστα. Δεν βλέπω κάποιον άλλον στο Catch Ολοκληρώνουμε λοιπόν την ακρόαση και σας δίνουμε τρία λεπτά για να συνοψίσετε. Η ελπίδα όλων μας είναι να δημιουργήσουμε δικαιοσύνη στην Ευρώπη ε, και ε, να υπάρχει ένας φίλος των πολιτών ικανός ε, να τον ακολουθήσει και σε αυτή τη διαδικασία που είναι και διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, γιατί θέλουμε οι πολίτες όλοι, όλα τα όργανα οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αισθάνονται ότι όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στην υπηρεσία τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβετε την απόφασή σας διαβάζοντας τα βιογραφικά, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία του διαμεσολαβητή, γιατί ας πούμε δεν είναι δυνατόν ο διαμεσολαβητής ε, να βρίσκεται ταυτόχρονα, να είναι ταυτόχρονα και μέλος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου μιας πολυεθνικής. Δεν συνάδει αυτό με την ε, εικόνα του διαμεσολαβητή. Ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής είναι κάποιος που επί πέντε χρόνια θα ακολουθήσει, θα παρακολουθήσει την εξέλιξη ε, των διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως θα πρέπει ε, να ξεκαθαρίζει και τις σχέσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και τα άλλα όργανα. Ο διαμεσολαβητής ε, είναι ακριβώς το καλύτερο εργαλείο που έχετε στην, διάθεσή σας έτσι ώστε να είναι αρρωγός στην καθημερινή σας εργασία και να ε, προωθήσετε την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φορτουνάτο, λέει η Πρόεδρος. Εμείς εδώ στην Επιτροπή Αναφορών είμαστε πάντα στη διάθεση των υποψηφίων. 11 και 20 έχει προβλεφθεί η επόμενη ακρόαση και επομένως ε, θα διακόψουμε τις εργασίες μας για 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Bueno, continuamos, continuo Λοιπόν, συνεχίζουμε, συνεχίζω στα ισπανικά. Είμαστε τώρα στην ακρόαση τη δεύτερη υποψήφια. Όπω ξέρετε, κάνουμε με αλφαβητική σειρά τι ακροάσει και τώρα λοιπόν είμαστε στην κυρία Τζούλια Λαφράντ. Λειτουργεί η μετάφραση. share. Um, um, which one do you want? English or do you want your language? If you want your Αγγλικά ή τη γλώσσα σας. Τα αγγλικά είναι στο 2. Νομίζω ότι έχουμε διαρμηνία και στη γλώσσα σας. Δεν ξέρω το. Τα εστονικά. Δεν τα βλέπω. 13. Το 13. Okay. Thank you very much. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά και από εκεί και πέρα θα περάσουμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να παρουσιάσω τις ιδέες μου για τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε όλη μου τη ζωή τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αξιοπρέπεια και το κράτος δικαίου ήταν πάντα πάρα πολύ, ήταν πάντα πάρα σημαντικά για εμένα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο σοβιτικό καθεστώς της Εστονίας και βίωσα από πρώτο χέρι τι σημαίνει να αποκτάς την ελευθερία και μετά να γίνεσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ε, ανέκτησε την ανεξαρτησία στη Εστονία, είχα την ευκαιρία να ζήσω και να σπουδάσω στο εξωτερικό. Σπούδασα ε, νομική στη Γερμανία, έμεινα στη Γαλλία και έμαθα αρκετέ ε, ξένε γλώσσε. Τα τρία μου παιδιά είναι εστονική και γαλλικής υπηκότητα. Οπότε είμαι ένα τέλειο παράδειγμα για το τι προσέφερε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην γενιά του Εράσμου. Είμαι Ευρωπαία. Αλλά δεν έχω ξεχάσει τις ρίζες μου που είναι από ένα μικρό νησί ψαράδων στην Εστονία. Τα μέλη της κοινότητας τώρα με παρακολουθούν και με ρωτάνε τι είναι αυτός ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής, τι κάνει. Και θα τους πω πώς βλέπω εγώ τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Θα σου το εξηγήσω και αν έχουν προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Διοίκηση, ο Ευρωπαίος δημοσιολαβητή εκεί για να τους βοηθήσει. Θα τους πω ότι έχουν θεμελιώδες δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν στον Ευρωπαίο Δημοσιολαβητή και ότι αυτός είναι ο θεματοφύλακας τη χρηστή διοίκηση και υπερασπιστή των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο Ευρωπαίο Δημοσιολογητή δεν θα πρέπει να κάνει έρευνες ή να επικαλύπτει το πολιτικό έργο των ε, Επιτροπών του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν πρέπει να επικαλύπτει ε, το έργο των διεθνών ε, οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης δεν είναι δικαστήριο. Δεν πρέπει να ακολουθεί τα πολιτικά του ή άλλα ένστικτα. Πρέπει να βασίζει τη δουλειά του στην καλή γνώση του νόμου αλλά και την ε, έννοια της δικαιοσύνης. Και αυτά έχω να σας προσφέρω γιατί είμαι δικηγόρος στο επάγγελμα. Έχω εμπειρία 15 χρόνια στο δικαστήριο της Εστονίας σε διοικητικά και συνταγματικά θέματα και τώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο ε, Στρασβούργο που είναι η συνείδηση της Ευρώπης. Διαχειρίστηκα πολλές υποθέσεις ε, για τρομοκρατία, περιβάλλον, γεωργία, απαγωγή παιδιών, ε, ελευθερία έκφρασης. Είχα επίση το θάρρος να ε, εκφράσω την αντίθεσή μου σε αμφιλεγόμενα θέματα, σε θέματα ζωής και θανάτου. Ξέρω τα προβλήματα των ανθρώπων πολύ καλά, αλλά γνωρίζω εξίσου καλά και την διοίκηση, γιατί υπήρξα δημόσιο υπάλληλο στην Εστονία, μια χώρα με ηλεκτρονική διοίκηση. Και ξέρω, ότι Ευρωπαϊκή, ε, ξέρω επίσης και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία πάρα πολύ καλά, γιατί ήμουν καθηγήτρια Ευρωπαϊκού Νόμου στο Πανεπιστήμιο του Τούρκου, του Τάρτου. Οι διεθνείς οργανισμοί μου έδωσαν λοιπόν την ε, αυτοπεποίθηση να μπορώ να σταθώ σε διεθνή σκηνικά. Ξέρουμε η δημοκρατία τι μπορεί να κάνει για τους πολίτες και δεν ήμουν ποτέ ε, φιλικά προσκύμενη σε συγκεκριμένο κόμμα, σε συγκεκριμένη παράταξη. Γι' αυτό, γι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει ο διαμεσολαβητής να είναι ε, να λειτουργεί με διαφάνεια, να είναι μερόληπτο για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ποιο είναι ο λόγο που είμαι υποψήφια σήμερα. Είμαι υποψήφια για το αξίωμα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, γιατί πιστεύω ε, στεναρά στη δυναμική του, στο τι μπορεί να κάνει για το καλό των ε, πολιτών. Γιατί γνωρίζω και είμαι εξοικειωμένη με την ισχύ που έχει αυτός ο ρόλος και ποια είναι επίσης τα προβλήματα. Και θα ήθελα να ενισχύσω ε, αυτή, τη, αυτά τα θετικά, σημεία και να επιλύσω τα προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα είναι ίσως ότι ε, οι, ευρωπαϊκοί, Ευρωπαίοι πολίτες έχουν ε, και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή γιατί οι συστάσεις του πλέον δεν βασίζονται στην ομοθεσία και οι θεσμοί σε πολύ σημαντικές υποθέσεις δεν δέχτηκαν τις συστάσεις του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Ένα παράδειγμα, το παράδειγμα που αφορά τις δαπάνες των μελών του Ευρωκοινοβουλίου, όπου το Ευρωκοινοβούλιο επέκρινε τον διαμεσολαβητή που δημοσιοποίησε το θέμα προτού να ακούσει την άποψή του. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, δίκαιη κρίση. Βλέπουμε επίσης ότι το ποσοστό των ε, ε, καταγγελιών έχει μειωθεί και ξέρω από τις στατιστικές ότι παρόλο που έχουμε πάνω από 500 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν μόνο 2.000 καταγγελίες ε, ετησίως ε, στο, Ευρωπα... Γραφείο του Ευρωπαϊκού Δημοσιολαβητή. Συζήτησα με δύο πρώην διαμεσολαβητές που αποτελούν πηγή έμπνευσης για την υποψηφιότητά μου και μίλησα σε πάρα πολλούς εθνικούς διαμεσολαβητές όπως και το Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς ε, Ινστιτούτου για τη Διαμεσολάβηση. Πολλοί από αυτούς είναι δικηγόροι και δικαστές. Και έχω ένα πολύ ξεκάθαρο όραμα για το γραφείο του διαμεσολαβητή. Και το όραμα αυτό είναι να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες της Ευρώπης, βασιζόμενοι σε δύο πυλώνες εμπειρογνωμοσύνη και γνώση και αίσθηση της δημοκρατίας και ανθρώπινη προσέγγιση. Και έχω ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο για το πώς θα το κάνω αυτό. Έχω ένα σχέδιο δράσης λοιπόν, σήμερα που το ετοίμασα για εσάς. Δεν έχω όμως αρκετό χρόνο για να μπω σε λεπτομέρειες. Μπορώ όμως να ε, επισημάνω πέντε σημαντικά σημεία. Πρώτον, οι καταγγελίες θεωρώ ότι θα πρέπει να ακολουθεί όλες τις διαμαρτυρίες και θα πρέπει να τις λαμβάνει όλες σοβαρά υπόψη, γιατί όλες δείχνουν ότι κάτι δεν είναι σωστό στην Ευρώπη. Κάθε διαμαρτυρία θα πρέπει να είναι ίση με την άλλη. Επίσης είναι σημαντικό να πιστεύουμε τους ευάλωτους, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τις μειονότητες, τους ετούντες άσυλο, τους πρόσφυγες που ζουν στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα άτομα με αναπηρία. Και θα σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία και τα δικαιώματα τους πρέπει να είναι σεβαστά. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό ε, έργο είναι η έρευνη της ίδιας πρωτοβουλίας προς όφελος των πολιτών και η πρώτη μου έρευνα θα έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση και την χρήση της τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση για να δω κατά πόσο είναι σύμφωνη με τα ε, δικαιώματα των πολιτών και τις ηθικές ε, αρχές. Επίσης, θα διερευνήσω πώς ε, μπορούν να συμμετέχουν τα άτομα με αναπηρία σε νομοθετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Και έτσι περνάω στο τρίτο σημείο, έχω σκοπό να συμμετέχω στις ε, δημόσιες διαβουλεύσεις της Επιτροπής όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών. Και σας διαβεβαιώνω ότι θα συμμετέχω ενεργά στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κωδικοποίηση της ε, ε, Ευρωπαϊκής Δομοθεσίας. Τέταρτη σημαντική παραμετρός είναι το να υπάρχει πρόσβαση για όλους τους πολίτες στο γραφείο, γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Δεν υπάρχει ένα δημόσιο αρχείο εγγράφων σε ένα, ε, οργανισμό που προωθεί τη διαφάνεια. Και αυτό θα το πράξω όσον αφορά τη διαφάνεια. Θα εργαστώ σε θέματα διαφάνειας από κοινού με εθνικούς διαμεσολαβητές. Και θεωρώ ότι πρέπει να προωθήσουμε μια κουλτούρα ανοιχτής ε, διοίκηση. και αυτό με φέρνει στο πέμπτο σημείο που έχει να κάνει με το συντονισμό και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκεκριμένα με την Επιτροπή Αναφόρων αλλά και με άλλες ε, ε, επιτροπές, ώστε να υπάρχουν μόνιμα, μόνιμη διεύλη επικοινωνία με του εθνικού διαμεσολαβητέ. σε θέματα όπως είναι η προστασία των whistleblowers. Κυρίες και κύριοι, θα είμαι ηγέτης με και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου ώστε να εργαστούμε αποτελεσματικά με πραγματικό αντίκτυπο και με ορατότητα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές προκλήσεις και θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται και ότι υπάρχει κράτος δικαίου. Οι επαφές μαζί σας και η υποστήριξη που είχα από εσά, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, και οι εμπνευσμένες συζητήσεις που είχαμε και υποστήριξη από διαφορετικά κρατημέλη και διαφορετικά κόμματα δείχνουν ότι συμφωνείτε μαζί μου. Και είναι πλέον καιρός να έχουμε έναν δικηγόρο, νομικό μάλλον, ως Ευρωπαίο διαμεσολαβητή. Θα είμαι η φωνή των Ευρωπαίων πολιτών και θα χρησιμοποιήσω τη γνώση μου και την εμπειρία μου ε, ε, για να σας υπηρετήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, we start with EPP and has... Ξεκινούμε με το ΕΛΚ. Ο Άξελ Βός έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μάλλον πρέπει λίγο να περιμένω. Ναι, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Λεφρανκ, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Θα είμαι σύντομος. Θέλω να μας εξηγήσετε το σχέδιο δράσης σας, να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα για να δούμε πώς μπορούμε να το κρίνουμε και επίσης μια επιπρόσθετη ερώτηση. Τι περιπτώσεις είχατε στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα ήταν πολύ σημαντικό να το μάθουμε και αυτό σε αυτή, αυτή τη στιγμή. Ναι, ευχαριστώ. Αυτό το πρόγραμμα δράση είναι πολύ συγκεκριμένο. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι η προσέγγιση του διαμεσολαβητή προς τους πολίτες, ώστε να είναι απλουστευμένη η πρόσβασή τους, να υπάρχει δυνατότητα χρήση των παραδοσιακών ε, ε, ε, αλλά και των ηλεκτρονικών διάβλων επικοινωνίας. Επίσης, μια έμφαση στην πολυπολιτισμικότητα, στην πολυγλωσία και επίσης να μπορεί ο διαμεσολαβητής να έχει live chat online, ζωντανή ε, συζήτηση με τους ε, πολίτες, επίσης ε, συνεργασία με τους εθνικούς διαμεσολαβητές και έχω και ακόμα μια ιδέα να υπάρχει απόσπαση ε, των εθνικών διαμεσολαβητών ε, στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή. Έχω συγκεκριμένε ε, ε, προτάσεις για τις ε, on initiative inquiries και ακόμα κάτι που θέλω να τονίσω είναι ότι Όλες οι υπηρεσίε που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των πολιτών, θα τι επισκεφτώ όλες τις υπηρεσίε αυτές. Όταν ξεκίνησα, στο δικαστήριο υπήρξαν 100.000 ε, υποθέσεις εκκρεμή περίπου, αλλά μπορώ να θυμηθώ δύο πολύ σημαντικές. Η πρώτη είχε να κάνει με την ομοιρία στην Ρωσία, με την υπόθεση ομοιρία στη Ρωσία. όπου καταλάβαμε ότι η καθημερινή χρήση βίας στους ομήρους οδήγησε φυσικά στην παραβίαση της συνθήκης, της Συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είχαμε πολλά θέματα εκεί, είχαμε γονείς που είχαν χάσει τα παιδιά τους αυτή την ε, τρομοκρατική επίθεση, οι οποίοι αυτοί ήταν παρόντες στην αίθουσα ακροάσεων. Και όταν ε, ανακοινώθηκε η απόφαση, οι καταγγέλλοντες είπαν ότι επιτέλους αποδόθηκε η δικαιοσύνη. Μία από τις πιο βασικές υποθέσεις ήταν αυτή. Υπάρχουν βέβαια και άλλες. Μια δεύτερη υπόθεση είναι το freedom of expression, ελευθερία έκφρασης, ρητορική μίσους σε ανώνυμα σχόλια στην Εστονία έλαβε χώρα αυτό και ασχολήθηκα και με αυτό και ήταν, ε, ήταν ε, μια θεμελιώδης αυτή η απόφαση για την ε, απαγόρευση της ρητορικής τους μίσους σε ανώνυμα σχόλια στο ίντερνετ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο κύριος Άμεριξ από το S&D. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ. Εμένα με πείσατε με τα όσα είπατε στην αρχική σας παρέμβαση, αλλά θα ήθελα να θέσω την ίδια ερώτηση που έθεσα και στον προηγούμενο υποψήφιο. Ο ρόλο του διαμεσολαβητή είναι κάτι παραπάνω από ε, νομικού διαμεσολαβητή. Είπατε δύο πράγματα γι' αυτό. Ποιοι είναι οι τρει συγκεκριμένοι στόχοι σα, τους οποίου δεσμεύεστε να επιτύχετε στη διάρκεια τη θητεία σα και ποια είναι οι τρει βασικοί τομεί. τις οποίους θέλετε να αντιμετωπίσετε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Κοιτάξτε, ε, είναι σαν να ξεκινάς ε, να τρέχεις. Θα πρέπει δηλαδή να μπει σε καλή θέση έτσι ώστε να τελειώσεις πρώτος ε, ή αν θες και να τελειώσεις τον αγώνα. Εγώ βλέπω λοιπόν τον νόμο ε, και το, το νομικό σύστημα σαν ένα καλό σημείο εκκίνησης. Είναι το βασικό εφόδιο που πρέπει να έχεις για να ξεκινήσεις ε, το τρέξιμο και μετά βέβαια για να μπορέσει να συνεχίσεις το τρέξιμο πρέπει να έχεις συνέστηση, πρέπει να είσαι αποτελεσματικός ε, και να έχει και όραμα. Το όραμά μου είναι ε, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής να προσεγγίσει, να έρθει πιο κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη. Είναι σημαντικό ε, να υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Διαμεσολαβητή από πλευρά των πολιτών, έτσι ώστε να βοηθηθούν οι πολίτες, αλλά να βοηθηθούν και τα όργανα, να η διοίκηση δηλαδή. Αυτό είναι το κεντρικό στοιχείο ε, ο κεντρικός μου πρώτος στόχος. Θα πρέπει ο διαμεσολαβητής να βγει από αυτή τη φούσκα ε, των Βρυξελών και να προσεγγίσει και τους ε, συνηγόρους του πολίτη στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να γνωρίζει και πώς αντιμετωπίζονται κάποια θέματα από τα νομικά συστήματα των χωρών. και Ακριβώς αυτό είναι το συγκλονιστικό ε, με τον διαμεσολαβητή. Βεβαίως ε, η δουλειά του θα βασιστεί στις ε, καταγγελίες αλλά κυρίως θα βοηθηθεί και από τις δικαιοδοσίες ίδιας πρωτοβουλίας που έχει. Όπως είπα και στο σχέδιο δράσης μου, εγώ θέλω να είμαι κοντά στους πολίτες, θέλω ε, να ε, είμαι βεβαία ότι οι καταγγελίες γίνονται δεκτές από τις ε, υπηρεσίες και ότι θα υπάρξει καλή διοίκηση. Έχω και ένα όραμα για το μέλλον γιατί ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής θα είναι αυτός Ε, ε, ο οποίος θα προωθήσει και τα θέματα που σχετίζονται με την ε, σύμβαση για τους ανθρώπους με αναπηρία. Η κυρία Μίλ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Λεφράνκ. Ο ρόλος του διαμεσολαβητή είναι ανεξάρτητος, όμως υπάρχει μια στενή σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη σαφήνεια μας ε, εξήγησατε τις αρμοδιότητες σας και πόσο σημαντική είναι για σας η ανεξαρτησία του διαμεσολαβητή. Γι' αυτό θέλω να σας συγχαρώ. Θα ήθελα να μάθω πιο ακριβώς ποιο θα είναι το πρόγραμμά σας, οι προτεραιότητές σας και ιδιαίτερα για την ίδια πρωτοβουλία που θα αναλάβετε. Θα κάνετε έρευνες συγκεκριμένες, έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις ή προθέσεις. Θα ήταν πολύ σημαντικό να μας τις παρουσιάσετε εδώ. Ευχαριστώ πως ε, υπόθηκε. Ο βασικός ρόλος είναι η επίλυση των ε, υποθέσεων, των καταγγελιών, αλλά Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να μείνουν ανώνυμοι από τους καταγγέλλοντες. Ε, υπάρχουν και διαμαρτυρίες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Υπάρχουν ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τα ταμεία, τα ευρωπαϊκά, τις υπηρεσίες. Άρα θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικοί με τις αρχές αυτές αλλά γενικότερα μπορεί να διακρίνει κανείς το ρόλο αυτό, ποια είναι τα γενικότερα προβλήματα που υπάρχουν και έτσι μπορεί να προβεί σε ε, προτάσεις ίδιας πρωτοβουλίας. Θα πρέπει να είμαστε όμως αποτελεσματικοί και γι' αυτό χρειάζεται έρευνα σε βάθος, ε, σε βάθος ανάλυση και επίσης να είμαστε δραστήριοι και ενεργοί στην ε, δημόσια διαβούλευση για νομοθετικές προτάσεις. Μπορεί ο Ευρωπαϊκός Δημοσιολογητής να κάνει προτάσεις και, για, και στην νομοθετική διαδικασία. Συνεργάζεται με το Ευρωκοινοβούλιο, με την Επιτροπή Αναφορών, που είναι μέλος η Επιτροπή ε, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο συνηγόρων του πολίτη. Άρα βλέπω τα own initiative inquiries έναν ιδιαίτερο ε, ρόλο, ένα ιδιαίτερο εργαλείο μάλλον για τον ε, διαμεσολευτή για να δει και να διακρίνει, να καταλάβει ποια είναι η χρηστή διαχείριση, να εντοπίσει τα λάθη στη διοίκηση ώστε να τα βελτιώσει. Γιατί όταν κάνει λόγο για κάτι το οποίο δεν εμπίπτει στις αρμοδιαίτητες του, τότε χάνει την αξιοπιστία του, τη φήμη του και φυσικά αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ε, να έχει εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των θεσμικών οργάνων. Έχω αναφέρει τις συγκεκριμένες προτάσεις στην ομιλία μου και τις έχω συμπεριλάβει και σε αυτό το πρόγραμμα δράσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you for green. Ευχαριστώ η κυρία Όκεν για τους πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ ε, που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Με εξέπληξε όταν είπατε ότι χρειαζόμαστε ένα νομικό. Νομίζω ότι ε, δεν χρειάζεται να είναι νομικό. προβλέπεται στον κανονισμό. Χρειάζεται να υπάρχει νομική βάση, νομικό υπόβαθρο στο γραφείο του διαμεσολαβητή και δεν χρειάζεται να είναι κάποιο νομική. Εγώ ε, έκανα δουλειά διαμεσολαβητή για 33 χρόνια στη Δανία, πριν ε, έρθω εδώ για 15 χρόνια και παρά το γεγονό ότι είχαμε εξαιρετικούς νομικούς, ε, δώσαμε ιδιαίτερη υποστήριξη στην Έμιλιο Ράιλι και ακόμα την υποστηρίζουμε. Και νομίζω ότι όσον αφορά τα θέματα εμπιστοσύνης, δεν ξέρω που το βρήκατε αυτό. Αν ε, νομίζω ότι θα αναλάβετε υποθέσεις όπου απλώς τα θεσμικά όργανα στο τέλος θα υποκλίνονται και θα λένε να προχωρήσουμε, τότε δεν κάνετε πραγματική δουλειά διαμεσολαβητή, διότι κάποιες υποθέσεις είναι πολύ δύσκολο να τις αναλάβει κάποιος και δεν έχετε τα μέσα ε, να λέσετε απαραίτητα ένα πρόβλημα. Θα πρέπει να το διαχειριστείτε και να βρείτε τρόπο να το διαχειριστείτε και δεν καταλαβαίνω και τι λέτε όταν μας λέτε ότι υπάρχει νομική βάση για το έργο εκεί. Πραγματικά με εκπλήσει αυτό. Αυτό το οποίο θα ρωτήσω εδώ είναι αν θεωρείτε ότι είπατε ότι θα είστε ότι φροντίστε να αναλαμβάνετε εκθέσεις πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι αυτή η οποία υπεκρίθηκε περισσότερο, η έκθεση Σελμάιερ, στηρίχθηκε πάνω από το 50% του Κοινοβουλίου και επιβεβαιώθηκε και στην ετήσια έκθεσή μας. Υπήρχε μεγάλη πλειοψηφία στην ετήσια έκθεση που υπερψήφισε την έκθεση. Ε, και ξέρετε ότι υπάρχουν καταγγελίες και τα ξέρετε αυτά, η υπόθεση Σελμάιερ, η υπόθεση Μπαρόζο, βασίστηκε σε καταγγελίες. Θα αναλάβετε εσείς τέτοιες υποθέσεις αν οριστείτε διαμεσολαβητής ή θα αναλάβετε μόνο εκθέσεις πρωτοβουλίες όπου θα είστε βέβαιοι ότι θα έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Είστε κατά τη έκθεση για τη διαφάνεια στο Συμβούλιο, η οποία θα χρειαστεί βέβαια πάρα πολύ χρόνο πριν καταλήξουμε στο αποτέλεσμα. Κύριε Άουκεν, τελειώνει ο χρόνος σας. Ορισμένες φορές είναι πολλές κατηγορίες και το Κοινοβούλιο ρωτήθηκε για το θέμα των επιδομάτων, γιατί ε, έχει γίνει και έρευνα στο παρελθόν για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι χρειάζεται τουλάχιστον 10 λεπτά για να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις, αλλά θα απαντήσω πολύ εύκολα σε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να είμαι σαφής. Δεν είναι δική μου ιδέα ότι ένα δικαστή είναι καλό για τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Είναι δική σα ιδέα, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι προβλέπεται στο καθεστώ του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, στο άρθρο 6, παράγραφο 2, που λέει ότι τα άτομα τα οποία είναι ικανά να αναλάβουν τα ανώτατα δικαστικά αξιώματα στη ε, χώρα τους, είναι ιδανικοί υποψήφοι για διαμεσολαβητές και δεν χρειάζεται να αποδείξουν ότι εργάζονται ως διαμεσολαβητές ε, κάπου αλλού στο παρελθόν. Αυτή είναι η επιθυμία του νομοθέτη και αυτό έγινε όταν εγκρίθηκε το καθεστώ του διαμεσολαβητή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το θεωρώ ότι αυτό γίνεται λόγω τη αμεροληψία και τη ανεξαρτησία και λόγω της δίκαιας διαδικασίας που είναι στο DNA των δικαστών. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι δικαστής απαραίτητος ο διαμεσολαβητή, Το είπα και αυτό και στην παρέμβασή μου. Και δεν σημαίνει ότι πάντα ο Ευρωπαίο Μεσολαβητής πρέπει να είναι δικαστής, αλλά αν έχετε υποψήφιο που είναι δικαστής με νομικές γνώσεις και ένας ανθρώπινο πρόσωπο και όλη την υπόλοιπη εμπειρία που χρειάζεται για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό σημείο κίνηση και είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβετε υπόψη και φυσικά εγώ ε, παραπέμπω στην συλλογική σα ε, σοφία επί του θέματο. Όσον αφορά τι έρευνε ίδια πρωτοβουλία, όπω σα είπα, πρέπει να γίνονται με σοφροσύνη. Διότι ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν θα πρέπει να αναλαμβάνει Καταγγελίε από πολιτικέ αντιπροσωπείε ή πολιτικέ ομάδε. Μόλι ξεκινήσει να κάνει κάτι τέτοιο Ευρωπαίος διαμεσολαβητή, θεωρείται φιλικά προσκύμενο σε κάποιε ε, ιδέε και δεν θα πρέπει να ισχύει κάτι τέτοιο, διότι κάθε πολίτη και κάθε θεσμικό όργανο πρέπει να εμπιστεύεται τον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή και πρέπει να διαβουλεύεται και με τα θεσμικά όργανα και να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα της ε, δίκαιης ε, δίκης πριν φτάσουν οι έρευνε τη ίδια πρωτοβουλία μέχρι τέλου. Και αυτό μπορώ να σα το ε, προσφέρω. Επιμονή, επιμονή και σεβασμό. Όπω είπε ο Γκίνσπουργκ, ανώτατο δικαστή στο Ηνωμένε Πολιτείε, έχω το θάρρο να κάνω αυτό στο οποίο πιστεύω. Και το στένο σημαίνει ότι θα πρέπει να καθοδηγήσω και τους υπολείπους να ε, μου συμπαρασταθούν και να σταθούν δίπλα μου από αυτό. Πρέπει να βασίζομαι σε πάρα πολύ καλή νομική γνώση. Ίσως θα είχα κάνει κάποια πράγματα διαφορετικά, δεν θα είχα σχολιάσει συγκεκριμένε περιπτώσεις, ε, ε, αλλά πριν ε, εμβαθύνω σε αυτά τα θέματα, σίγουρα θα είχα συζητήσει με τα συμβαλώμενα μέρη και βάσει και τις επιχειρηματολογίες μου και θα είχα βασίσει ε, τα επιχειρήματα σε ό,τι έχουν να πούνε τα θεσμικά όργανα, ώστε να πει κάποιο ότι Α, αυτό μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και θα ρωτήσω εγώ γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αν ρωτήσω γιατί, θα πρέπει αμέσω να με εξηγήσουν γιατί δεν μπορούν να το κάνουν και αν πούνε ότι είναι λόγω νομοθεσία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με το ψήφισμα και τη σύσταση και το Κοινοβούλιο είναι εδώ για να μα βοηθήσει. Ο Ευρωπαίο Δημοσιολαβητή είναι ο σύνδεσμο τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Thank you. Now, e Ευχαριστώ πολύ, Ισιάρα και ο Καλή σας ημέρα και καλώς ορίσατε. Θα ήθελα να σας υποβάλω αρκετά ερωτήματα ε, από δύο πεδία στην ουσία. Το πρώτο είναι το lobbying ε, στα ευρωπαϊκά όργανα. Πιστεύετε ότι οι κανονισμοί για το λόμπι και για ε, τις ε, δημόσιες και ιδιωτικές διαδικασίες είναι σωστές και αν όχι, τι πρέπει να αλλάξει. Δεύτερη ερώτηση, το ρώτησαν και άλλοι, αλλά δεν απαντήθηκε κανονικά. Πιστεύετε ότι οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης ε, των νομοθετικών πράξεων μέσω τριμερών διαλόγων είναι διαφανείς διαδικασίες για τους πολίτες και αν όχι τι πρέπει να αλλάξει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βουλευτά για αυτό το ερώτημα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Πολλά ε, πρέπει να γίνουν ακόμα όσον αφορά το lobbying τις ομάδες άσκησης πίεσης. Ε, πρέπει να ε, είναι ε, υπόλογες οι ομάδες lobbying, πρέπει να υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες και οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει μητρό διοργανικό για όλες τις ομάδες πίεσης και οπωσδήποτε ο Ombudsman έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί το μητρό αυτό και τον με τον οποίο συμπεριφέρονται οι ομάδες πίεσης. Βεβαίως αυτά θα πρέπει να γίνουν ε, βήμα προς βήμα ε, έτσι ώστε να καλλιεργήσουμε και την κουλτούρα της ανοιχτής διαπραγμάτευσης. Ε, συγγνώμη, διακυβέρνησης. Όσον αφορά τις διαδικασίες, θα πρέπει και οι πολίτες να έχουν την ε, δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εργασίες της Κομισιόν, να δουν αν ακολουθούνται οι σωστές διαδικασίες. Αυτό αφορά την εφαρμογή του ε, Ευρωπαϊκού Νόμου στις χώρες μέλη. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος όμως της ερώτησής σας, πιστεύω ότι στους τριμερείς διαλόγους είναι σημαντικό να επανερχόμαστε στα κράτη-μέλη και να ξαναδούμε τον ρόλο των κρατών μελών και νομίζω ότι είναι σημαντικό να δουλέψουμε ε, και να συνεργαστούμε και με τους ε, εθνικούς διαμεσολαβητές γιατί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, στην προσπάθειά του να ε, διαλευκάνει τα προβλήματα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση ε, θα πρέπει να έχει την αρρωγή των εθνικών διαμεσολαβητών που οπωσδήποτε μπορεί να λέει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πρωτοβουλίες, οι νομοθετικές πρωτοβουλίες στις διάφορες διάφορες επιμέρους χώρους. Χώρες. Ε, και βεβαίως θα πρέπει να διασφαλίζει ή να ελέγχει το κατά πόσο υπάρχει διαφάνεια και προσπελασιμότητα. Δεν βλέπονται εδώ τον κύριο Γεωργούλη της Γκουέ, άρα ξεκινάμε ε, τον δεύτερο γύρο. Υπενθυμίζω ένα ε, λεπτό η ερώτηση, ένα λεπτό η απάντηση. Ξεκινάμε με τον κύριο Βίνθε του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λεφράνκ που είστε εδώ. Νομίζω ότι μας δώσατε ε, μια πολύ λεπτομερή και ολοκληρωμένη παρουσίαση. Έχω όμως ε, ακόμα μια ερώτηση. Θυμάστε την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, είπατε ότι έχετε μεγάλη εμπειρία. Ε, πώς ε, μπορεί να σας βοηθήσει στην εργασία σας ε, η δική μας Επιτροπή. Είπατε στο πρόγραμμά σας ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να καλύπτονται από τον διαμεσολαβητή. Με ποιο τρόπο ακριβώς. Δεύτερον, όσον αφορά την επικοινωνία στο πρόγραμμά σας αναφέρεστε στην επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα τι γίνεται όσον αφορά την επικοινωνία με το κοινό. Γιατί εάν επικοινωνούμε καλύτερα με το κοινό, τότε θα έχουμε και περισσότερους ανθρώπους που θα έρχονται σε επαφή με τον διαμεσολαβητή. Πώς αυτό μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμά σας. Ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω στα εστονικά. Ε, Σεβόμενη την πολυγλωσία ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ε, είπα και προηγουμένως, οι ελευθερίες αποτελούν δικαιοδοσία του διαμεσολαβητή και επομένως είναι δικαίωμα των πολιτών να έρχονται σε επαφή με τον διαμεσολαβητή και βεβαίως πρέπει όντως να επικοινωνούμε περισσότερο με τους Ευρωπαίους πολίτες. Εάν δείτε το πρόγραμμά μου θα διαπιστώσετε ότι ε, ε, αναφέρομαι σε κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν ε, τουλάχιστον στην αρχή της ε, θητείας μου ε, συγκεκριμένα κάποιες επισκέψεις οι οποίες δεν είναι επισκέψεις αυροφροσύνης προς τους εθνικούς συνηγόρους του πολίτη. Θα μου δοθεί η ευκαιρία να συζητήσω και με τους συνηγόρους σε επίπεδο κρατών αλλά και με τον κόσμο. Πραγματικά αυτός θα πρέπει να είναι ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Έχω άλλη μια ερώτηση. Ο κ. έχει σχετικά με τις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, διαμεσολαβητή. Ε, σαν διαμεσολαβητής πιστεύετε ότι ο ρόλος σας είναι με ε, να προβλαβαίνετε ενδεχομένως ε, ε, σε μερικές περιπτώσεις ε, τα προβλήματα. Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, βλέπουν τα ευρωπαϊκά όργανα οι πολίτες. Πώς φαντάζεστε ότι μπορείτε να κλείσετε αυτές τις, αυτά τα κενά στην επικοινωνία και στην εμπιστοσύνη Ευχαριστώ που απάντησε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτό συνδέεται με τα όσα είπα απαντώντας την προηγούμενη ερώτηση, πιστεύω ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ε, ο διασύνδεσμος ανάμεσα στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και εδώ στην Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου ε, πραγματικά βρίσκεστε στην αιχμή του δόρατος. έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε αναφορές ε, σχετικά και με την εφαρμογή του νόμου στις ε, χώρες μέλη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ανοιχτός διαρκής διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στον Ευρωπαίο ε, Διαμεσολαβητή και της, την Επιτροπή Αναφορών. Πέρα δηλαδή από τις ετήσιες αναφορές, τις ετήσιες εκθέσεις, συγγνώμη, όσον αφορά την ε, της δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών θα πρέπει να υπάρχουν και πιο ε, καθημερινές ε, επαφές και ο δεσμός ανάμεσα στην Επιτροπή Αναφορών και τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολογητή θα πρέπει να ενισχυθεί. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βεντρέν, ξέρετε ότι η ομάδα Renew Europe είναι απολύτως δεσμευμένη στη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, όπου το, θα υπάρχει το εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου, το, της Κομισιόν, αλλά και των πολιτών. Ε, ο διαμεσολαβητής, όπως είπατε, παίζει σημαντικό ρόλο στον εκδημοκρατισμό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην συμπερίληψη των προβληματισμών των πολιτών ε, στο πρόγραμμα εργασίας. Ε, οι πολίτες περιμένουν περιμένουν βέβαια συγκεκριμένες δράσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα περιμένω να μου πείτε και την άποψή σας για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτή τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και τι μπορείτε να προτείνετε έτσι ώστε να είναι πιο ενεργή η συμμετοχή των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Επιτέλους μπορώ να μιλήσω και γαλλικά, μια γλώσσα που αγαπώ πολύ. Όταν έγινε η συντακτική συνέλευση υπό την ε, ηγεσία του Ζισκάρ Ντεστένς, ε, εγώ ήμουνα ε, μια νεαρή υπάλληλο του Υπουργείου Δικαιοσύνη τη Εστονία τότε. Δεν ήμασταν ακόμα μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είχαμε προσκληθεί ω χώρα πρώτη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήμασταν συνδεδεμένη χώρα και θυμάμαι πάρα πολύ καλά το περιβάλλον και θυμάμαι επίση ότι ήταν ο πρώτος Ευρωπαίος διαμεσολαβητής, ο οποίος ε, ε, είχε την ιδέα να συμπεριληφθεί το άρθρο 41 στη συνθήκη. είναι Ένα άρθρο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους γιατί αναφέρεστε στη χρηστή διαχείριση. Και ε, φυσικά χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία και πολύ θα ήθελα να συμμετάσχω ως ε, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής σε αυτή την πρωτοβουλία κάνοντας μια κοινή δήλωση με τους εθνικούς ε, διαμεσολαβητές, ε, διότι είναι πολύ σημαντικό να ακούσαμε και τη δική τους την άποψη, προκειμένου να υπάρχει πραγματικά ε, μια συνολική εικόνα για τις ανάγκες των πολιτών στις χώρες μας και όχι μόνο σε επίπεδο Βρυξελών ή Στρασβούργου. Και χαίρομαι που θα έχουμε και τα 25 χρόνια του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή την επόμενη χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπεχούμεα τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κυρία Λαφράνκ που βρίσκεστε εδώ και για τα όσα μας είπατε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τα fake news, ε, τις ψευδείς ειδήσει και τον αρνητικό αντίκτυο που έχουν στην ανοιχτή δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν οι εχθροί της ε, ανοιχτής δημοκρατίας, ε, αυταρχικά καθεστώτα, ε, και θα ήθελα να ξέρω πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τα fake news ε, και τι συγκεκριμένα μέτρα μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή προκειμένου να σταματήσει η χρήση των fake news και του αντίκτυπου που έχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την ερώτηση αυτή. Εξέφρασα ήδη ότι έχω εμπειρία στο θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Βεβαίω ε, και πάλι σα υπενθυμίζω και τι αρμοδιότητε του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή που ε, βρίσκεται εκεί για να φροντίσει να υπάρχει χρηστή διαχείριση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και φυσικά όταν υπάρχουν ρητορίε μίσου για τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή θα πρέπει να εξετάσει πώ μπορούν να λυθούν τα θέματα αυτά σε επίπεδο διοίκηση. Όσον αφορά την ρητορία μέσους και την εξάπλωση της ρητορίας μίσου στα κράτη-μέλη και των fake news, ε, εδώ και πάλι είναι θέμα συνεργασίας με τους εθνικούς ε, συνηγόρους του πολίτη σε, στο επίπεδο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μέστρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Λαφράνκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Μια αντίστοιχη ερώτηση που έκανα και στον προκάτοχό σας, τον προηγούμενο υποψήφιο. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει αυτή η απόσταση μεταξύ πολιτών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Εσείς αναφέρετε ότι είναι γραφειοκρατία. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό. Ε, πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε οι πολίτες να προσεγγίσουν περισσότερο τα θεσμικά όργανα. Εσείς αναφέρεστε στα chats ε, προηγουμένως, μία από τις προτάσεις για να μπορέσει κάποιος να προσεγγίσει καλύτερα τους πολίτες. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα να λύσει το θέμα αυτό ε, το μέτρο. Στην παρέμβασή σας στην αρχική ε, αναφερθήκατε σε αυτή την εικόνα σορα, σοβαρότητας. Θεωρείτε ότι το να κάνει τσάτ με τους πολίτες θα προσθέσει σοβαρότητα. Και επίσης ε, πώς μπορούμε να, να, κάνουμε, να φροντίσουμε οι πολίτες να νιώσουν ότι υπάρχει καλύτερη πρόσβαση και είμαστε πιο κοντά. Very much, member. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, ωραία ερώτηση. Είναι ακριβώ αυτό που χρειαζόμαστε για να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και να είμαστε παρόντες, να δείξουμε με την παρουσία μας ότι είμαστε εκεί και ότι νοιαζόμαστε. Είναι μια δυνατότητα να είμαστε προσβάσιμοι, να μην φοβούνται, να μας πούν τα προβλήματά τους. Ο καθένας που έχει καλή γνώση, αλλά και ένα ανθρώπινο πρόσωπο, μια αίσθηση δικαιοσύνης. Όταν τα διαθέτει όλα αυτά, δεν είναι εύκολο να τα επικοινωνήσει με μια απλή γλώσσα. Αυτό χρειάζονται οι πολίτες. Και ο άλλος ο λόγος είναι να είμαστε ορατοί όχι μόνο δημιουργώντας τίτλους ε, στις ειδήσει, αλλά μέσα από την δουλειά το έργο μας. Άρα ε, έχω σκοπό να δημοσιεύουμε σε εβδομαδιαία βάση τα βασικά, τις βασικές καταγγελίες που έχουν γίνει σε διαφορετικές γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό για τις συγκεκριμένε υποθέσεις και το αποτελεσματικό μας έργο. Και φυσικά να επισκεπτόμαστε και τα κράτη-μέλη. Κυρία Ντανούκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Λαφράνκ. Έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Σε ποια πλευρά είστε σε μια περίπτωση διαφωνίας ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μιλάμε για μια περίπτωση για τον κανονισμό που αφορά την αμοδιότητα του Ευρωπαίου Δημοσιολευτή, ένα έγγραφο που έλαβε το Κοινοβούλιο και ότι έχει το δικαίωμα ο Δημοσιολευτής να κάνει συστάσεις όταν θεωρεί ότι ο... το θεσμικό όργανο δεν, είναι... δεν λειτουργεί σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου, ότι δεν εφαρμόζει μάλλον την απόφαση του δικαστηρίου. Εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο αυτό, αλλά ε, υπέβαλαν ένσταση η Επιτροπή και το Συμβούλιο, οι νομικές υπηρεσίες τους, ε, με το εξή επιχείρημα. Σύμφωνα με το άρθρο 228 της Συνθήκης για την Κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι σε θέση ο διαμεσολευτής να υποβάλει ερωτήματα σε θέματα κακοδιοίκησης, υπό οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Δεν μας έχει δώσει απάντηση το Συμβούλιο, αλλά η νομική υπηρεσία έδωσε αυτή την γνώμη. Εσείς με ποιανού το μέρος είστε, του Ευρωκοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. Αρχικά να, να συγχαρώ το Κοινοβούλιο για την αναθεώρηση του ρόλου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, κάτι που δεν έχει γίνει μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία. Και αν μου κάνετε την τιμή να με εκλέξετε θα είμαι, να με, να με ουσιαστικά ο βασικός συνομιλητής για αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις και θα εκφράσω τις απόψεις μου. Θεωρώ ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολευτής έχει άλλους τρόπους να επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Διοίκηση και τα θεσμικά όργανα και αυτό ονομάζεται Ombuds Prudence, δικαιοδοσία του διαμεσολαβητή αυτό προκύπτει από αποφάσει του δικαστηρίου και θεωρώ ότι ο διαμεσολαβητή θα πρέπει να είναι παρόν για να δει ότι η διοίκηση ε, υιοθετεί τι σωστές αρχές. Δεν είναι ο ρόλος του να επιβλέπει την εφαρμογή των αποφάσεων άλλων οργάνων και θεσμών, αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση, χάρη, για αποφάσει του δικαστηρίου που δεν εφαρμόζονται από κράτη-μέλη, τότε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητή θα πρέπει να, ε, είναι, να εξασφαλίσει ότι αυτή η δικασία θα ακολουθήσει την, ε, το σωστό τρόπο διοίκηση. Ε, είναι λοιπόν, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του διαμεσολαβητή, όμως παράλληλα βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή γνώση της νομοθεσίας για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των θεσμών ε, και την εμπλοκή των πολιτών. Ευχαριστώ. Κύριε Λοτόφσκι. Όχι. Κύριος Κάρθιαν Φουρόρε δεν είναι παρόν, οπότε ξεκινάμε με τη δικασία Catch κυρία Εύριν και ο κύριος Κώσα ζήτησαν το λόγο. Με συγχωρείτε, δεν σας είδα. Έχετε το χρόνο σας. Χωρίς μικρόφωνο μιλητής. Okay. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας, ο κύριος Φουρόρε, εσείς επικρίνατε έρευνας οι οποίες έγιναν από την παρούσα διαμεσολαβήτρια, την κυρία Οράιλε, οι οποίες κατά την άποψή μου προσέδωσαν αξία στο ρόλο του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή αυτά τα χρόνια. Ε, προστασία των πολιτών και τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και διοντολογίας στα θεσμικά όργανα. Αναφέρομαι σε σημαντικές έρευνες που έκανε η παρούσα διαμεσολαβήτρια για την ε, κακή διαχείριση που αναφέρθηκε κατά τον ε, διορισμό του πρώην Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Μπαρόζο, ε, ο οποίος προσελήφθη πολύ σύντομα μετά την ε, θητεία του στη Goldman Sachs. Και επίσης ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Goldman Sachs είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος δρά με σκέους ε, σκοπούς και υπάρχουν και αντίστοιχα στοιχεία για τον ορισμό του Μάρτιν Σελμάγερ ως Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και έρχομαι στην ερώτησή μου. Εσείς ουσιαστικά θεωρείτε ότι δεν θα πρέπει να ακολουθούμε αυτή την οδό εάν εκλεγείτε. Ε, θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε αυτή την πτυχή σας παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αναφέρθηκα στις ε, επικρίσεις ε, που είχαν εκφραστεί ε, και στα ακαδημαϊκά έγγραφα και στον τύπο χωρίς εγώ να ασκήσω κριτική ή να επικρίνω. Το θέμα δεν είναι πώς ε, τα ίδια τα θέματα, αλλά πώς αντιμετωπίζει κανείς ε, τα θέματα και πώς διατηρεί την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, γιατί εάν ε, χαθεί ε, η υπόλοιψη των, ε, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, τότε θα πάψουν και οι καταγγελίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δίκαιες διαδικασίες και να γίνεται σεβαστή η δίκαιη δίκη. Το θέμα δεν είναι blaming and shaming συγκεκριμένων ανθρώπων, αλλά να αλλάξουν κάποια στοιχεία στις δομές και οπωσδήποτε να υπάρχει, όπως το είπατε και εσείς, συστηματικά διαφάνεια. Και ως δικηγόρος... Ε, αυτό ξέρω και αυτό θέλω να προωθήσω. Πιστεύω ότι πραγματικά ε, ε, θέλουν οι πολίτες έναν άνθρωπο στο πλάι τους που να τους πει πώς μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Δεν χρειάζονται κάποιους που απλώς θα γράφουν τους πηχιαίους τίτλους είναι καλό να στρέφεται κανείς ε, και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως, αλλά πρώτα απ' όλα ε, ε, χρειάζεται καλή προετοιμασία, καλή διαρεύνηση και οπωσδήποτε να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των πολιτών και όχι όλα τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι οι μικροί ψαράδες στο χωριό μου ίσως δεν ξέρουν καν τους ανθρώπους που μόλις αναφέρατε, αλλά θέλουν οπωσδήποτε καλή διοίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια διοίκηση που θα μπορούν να εμπιστεύονται. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε και το δεύτερο γύρο, τώρα ξεκινάμε ένα τρίτο γύρο, είναι Catch the Δύο έχουν ζητήσει το λόγο, η κυρία Εύρεν και ο κύριος Κώσα. Η κυρία Εύρεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα γαλλικά γιατί ξέρω κύριε Λιουφράγκ ότι τα γαλλικά σας είναι εξαιρετικά, τα κατανοείτε απολύτως και σας συγχαίρω γι' αυτό. Θα ήθελα να ζητήσω ε, συγγνώμη για την ε, ε, αργοπορία μου. Δυστυχώς ήμουν αποκλεισμένη σε ένα τρένο. Σύμφωνα με το τελευταίο βαρόμετρο, ξέρουμε πλέον ότι 45% των Ευρωπαίων πολιτών δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του ως Ευρωπαίους πολίτης και δεν γνωρίζει και την ύπαρξη ή τον ρόλο του Ευρωπαίου διαμεσολαβητή. Ε, δεν επανέρχομαι ε, στο γεγονός που αναφέρθηκε ήδη ε, ότι αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Πώς προς πώς προτίθεστε ε, να αλλάξετε ε, την κατάσταση, να γίνει πιο ορατός ο ρόλος του διαμεσολαβητή, να γνωρίσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους οι πολίτες και πώς να θα συνεργαστείτε με τους εθνικούς διαμεσολαβητές. Ε, νομίζω ότι αναφερθήκατε σε κάποια απόσπαση των Ευρωπαίων συγγνώμη, των συνηγόρων του πολίτη. Εγώ απήντησα ε, επανειλημμένα σε παρόμοια θέματα, ε, σε παρόμοιε ερωτήσεις. Ε, τα ανέφερα άλλωστε και στην προαρχική μου παρέμβαση. Βρισκόμαστε σήμερα στις 3 Δεκεμβρίου. Δεν μπορούμε να είμαστε δυσυπόστατοι. Εγώ θα ήθελα πολύ όμως να είμαι στο συνέδριο ε, που ξεκίνησε ο συνήγορος του πολίτη της Γαλλίας ε, σχετικά με τους ε, καταγγέλλοντες, τους whistleblowers. Πρέπει και για τέτοια θέματα να συνεργαστούμε με τους εθνικούς διαμεσολαβητές, τους συνηγόρους του πολίτη δηλαδή στις διάφορες χώρες οι εθνικοί <clears throat> διαμεσολαβητές μπορούν να ασχοληθούν ε, και με θέματα τα οποία μπορεί να είναι ευρωπαϊκού ε, ενδιαφέροντος ε, στη διάρκεια των διαφόρων συναντήσεων που είχα με εθνικούς διαμεσολαβητές διαμόρφωσα την εντύπωση ότι αυτή η συνεργασία μεταξύ δηλαδή Ευρωπαίου και Εθνικών Διαμεσολαβητών δεν είναι πολύ μεγάλη ε, τα είπα και προηγουμένως ε, σχετικά με την παρουσία ε, στα κράτη-μέλη. Είπα λοιπόν ότι η Ευρώπη ξεκινάει στα κράτη-μέλη. Επομένως οι επισκέψεις επιτόπου, οι συναντήσεις με τους συνηγόρους σε εθνικό επίπεδο και με τους πολίτες είναι ένα πρώτο βήμα απαραίτητο έτσι ώστε να προσεγγίσει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής τους πολίτες. Ο κύριος Κώσα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε ε, τον λόγο. Είμαι και εγώ δικηγόρος και κατανοώ πλήρως ε, την ε, ε, κατάσταση. Ίσως θα διαφωνήσω και με κάποιους συναδέλφους μου. Γιατί το να είναι κανείς δικηγόρος δεν μπορεί να είναι ούτε μειονέκτημα ούτε πλεονέκτημα, αλλά ως δικηγόρος μπορεί κανείς να έχει μεγάλη εμπειρία στον νομικό τομέα πόσα θα χρησιμοποιήσετε εσείς αυτή την εμπειρία σας έτσι ώστε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής να γίνει πιο αποτελεσματικά γνωστός σε όλη την Ευρώπη. Ε, δεν ξέρουν πολύ την, ε, το διαμεσολαβητή, δεν ξέρουν τη διαδικασία με την οποία μπορούν να υποβάλουν ε, κάποια καταγγελία. Θα ήθελα να μου πείτε τα σχέδιά σας για το θέμα αυτό. Το δεύτερο αφορά άτομα με αναπηρία. Υπέβαλε το ερώτημα αυτό και στον προηγούμενο υποψήφιο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το πρόγραμμά σας. Αναφέρατε ότι ε, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα ε, των ανθρώπων με αναπηρία είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πώς θα ελέγχετε όμως ε, την εφαρμογή αυτού, αυτής της σύμβασης. Ευχαριστώ πολύ ως απάντηση. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, κοιτάξτε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να καλούμε εθνικούς ε, συνηγόρους ε, στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έτσι ώστε να τον συνεπικουρούν σε ορισμένες περιπτώσεις γιατί και οι, και εθνικοί διαμεσολαβητές ε, θα ε, μπορούν να φέρουν στις χώρες τους την ευρωπαϊκή εμπειρία και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, θα κατανοεί το εθνικό περιβάλλον όπως είπατε ε, και προηγουμένως, ε, υπάρχουν άνθρωποι ε, οι οποίοι θέλουν να έχουν προσβασιμότητα και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, οι πολίτες, οι οποίοι δυσκολεύονται ή διστάζουν να έρθουν σε επαφή με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή γιατί νομίζουν ότι θα πρέπει να μιλάνε καλά αγγλικά ενώ έχουν δικαίωμα για μετάφραση κλπ. Επίσης, όσον αφορά ε, την ε, ε, σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τους ανθρώπους με αναπηρία, υπάρχει ένα πρωτόκολλο εθελοντικού προαιρετικό, εθελοντικού χαρακτήρα που δεν έχει ακόμα επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσε ας πούμε να είναι αυτό ένα πρώτο έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Ε, και βεβαίως ε, συχνές επαφές ε, με την Επιτροπή Επιτήρησης που βρίσκεται στη Γενέβη. Να πω επίσης ότι θα ήθελα να δημιουργήσω ένα focal point στο γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ακριβώς για τα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Όουκεν, τελευταία από τη διαδικασία Catch the Eye. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Παρ' όλα αυτά, η σύγχυση που έχω εξακολουθεί να υπάρχει. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και τους εθνικούς διαμεσολαβητές. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Επίσης, ε, για να πάει κανείς στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν μπορεί να το κάνει τόσο άμεσα, θα πρέπει να είναι σε μια οργάνωση κτλ. Είναι λίγο ε, απλοϊκό αυτό που κάνετε, να τους συγκρίνετε και να τους μπερδεύετε έτσι, δηλαδή τους τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή με τους εθνικούς διαμεσολαβητές ε, και προκαλεί κάποια σύγχυση. Να σας ρωτήσω λοιπόν στο άρθρο 6, ε, δεν το θυμάμαι ίσως καλά, πάντως ε, αναφέρεται στην ανεξαρτησία του ε, Ευρωπαίου Διαμισολαβητή και λέει ότι ο Διαμεσολαβητής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, τόσο ανεξάρτητος όσο ο δικαστής. Δηλαδή εδώ επιμένουμε στο ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι ε, ε, ανεξάρτητος ο διαμεσολαβητής σχετικά με την ανεξαρτησία ε, αναφέρεται το θέμα σε σύγκριση με τους δικαστές όχι γιατί ε, με την έννοια ότι είναι καλύτερος ένας διαμεσολαβητής που έχει υπάρξει δικαστής αλλά γιατί έχει δυνατότητα ανεξάρτητης διαρεύνησης. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που συμφωνούμε ότι πρέπει ο διαμεσολαβητής να είναι ανεξάρτητο και αμερόληπτος, πρέπει να είναι ηθικός και να αποφεύγει συγκρούσεις συμφερόντων. Και αυτό είναι και στην έκθεση τη Επιτροπή Αναφορών για την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Και πρέπει να θεωρείται και αμερόληπτος και ανεξάρτητο από του πολίτε. Επομένω, ε, πρέπει και να γίνονται αλλά και να φαίνονται έτσι. Επομένω, ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή δεν πρέπει να θεωρείται ότι έχει πολιτική επιρροή, διότι τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστία και σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστία με τα θεσμικά όργανα και ω δικαστή που έχω την αμεροληψία και την ανεξαρτησία στο DNA μου και δεν έχω πολιτική ε, φιλική, δεν είμαι φιλικά προσκύμενη σε κάποιο πολιτικό κόμμα, αυτό θα κάνω. Δεν θέλω να φαίνεται ότι ο διαμεσολαβητής είναι προκατηλημένος και, και δέχεται σήμερα προτάσεις από κάποιον και αύριο προτάσεις από κάποιον άλλον. Ο διαμεσολαβητής πρέπει να παραμείνει σταθερό στι ε, αρχέ του και στα του και σε αυτό που θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτε για το διαμεσολαβητή. Αλλά ο διαμεσολαβητή, και το είπα και σε μια συνάντηση με μια πολιτική ομάδα, δεν είναι και ο Άγιο Βασίλη, δεν είναι το χρυσόψαρο για το ψαρά που παίρνει τα ψάρια όλων, δεν μπορεί να είναι όμοιρο κανένα πολιτικού κόμματο ή καμία μη κυβερνητική οργάνωση, είναι εκεί να υπηρετεί του Ευρωπαίου πολίτε. Και αν συμφωνείτε μαζί μου, ελπίζω να έχετε και τη συλλογική σοφία να αποφασίσετε να έχετε έναν εξάρτητο και αμερόληπτο με διαμεσολαβητή που ξέρει πάρα πολύ καλά τα βασικά στοιχεία. Ε, και θυμάται από πού ξεκίνησε για να καταλήξει εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχετε λοιπόν το λόγο για τρία λεπτά για να ολοκληρώσουμε την ακρόασή σας. Ευχαριστώ πολύ τα μέλη και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ εξαιρετική ανταλλαγή ιδεών με πολύ έμπνευση. Σας ευχαριστώ πολύ και να τονίσω για άλλη μια φορά ότι ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής είναι ο δεσμός, σύνδεσμος ανάμεσα, ανάμεσα στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Δεν είναι δικαστήριο ούτε πολιτικός θεσμός, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά και στα δύο. Και αν με εκλέξετε θα ξέρετε ακριβώ τι να περιμένετε. Θα έχετε μια διαμεσολαβητή, η οποία θα είναι αμερόληπτη με τα κατάλληλα προσόντα επαγγελματίας που θα σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η οποία έχει το αίσθημα δικαιοσύνης και μια ανθρώπινη προσέγγιση όπως σας παρουσίασα πριν στο όραμά μου. Επίσης πρέπει να έχει μια σφαιρική εικόνα του τι συμβαίνει και ισορροπημένες ηθικές λύσεις. Δεν φοβάμαι να πω την αλήθεια για να εξασφαλίσω τη χρηστή διαχείριση. Θα εργαστώ με το κεφάλι, την καρδιά και με τα χέρια μου. Και θα επανέλθω τώρα στους ψαράδες. Θα μιλήσω στονικά. Οι ψαράδες λοιπόν, οι ναύτες ξέρουν ότι τα οι καυγάδε στη θάλασσα είναι πολύ άσχημοι, γιατί άμα μαλώσουμε κάποιο στη θάλασσα δεν μπορεί να κρυφτεί πουθενά. Και γι' αυτό επιλέγουν πολύ προσεκτικά ποιο θα πάρουν μαζί του οι ναύτε, οι ψαράδε. Ε, διαλέγουν αυτού που γνωρίζουν καλά τη δουλειά του, που είναι ισορροπημένοι, που δεν φοβούνται την ε, καταιγίδα και που είναι ψύχρεμοι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Τελειώσαμε αυτό το τμήμα. Ξεκινάμε στις 2.30 και μισή και πάλι έχουμε τρεις ακροάσεις. Να φάτε καλά.